Uh, if we can get ready to start, that would be great. Thank you. Right. Good afternoon, everyone. Καλό απόγευμα σε όλους. Το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη σήμερα το απόγευμα είναι οι κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησεις των κρατών μελών, ανταλλαγή απόψεων είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων χωρίς, εισηγητή, χωρίς, ε, συγγνώμη, χωρίς έκθεση νομίζω. Ε, δίνω το λόγο στον κύριο ε, Ρή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ναι, πράγματι δεν έχουμε έκθεση στα χέρια μας και σύμφωνα με το, χρονοδιάγραμμα που ενέκριναν οι συντονιστές, ε, την Τρίτη θα μπορέσουμε να υποβάλουμε στους ε, μεταφραστές το κείμενο, ώστε στις 17 στην έκτακτη συνεδρίαση να έχουμε αντίγραφο της ε, μεταφρασμένης έκθεσης. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να συζητήσουμε την ανακοίνωση της Κομισιόν, δηλαδή την πρόταση της Κομισιόν, για απόφαση του Συμβουλίου που σύμφωνα με την ε, διαδικασία της συναπόφασης θα πρέπει να σχολιαστεί από το Κοινοβούλιο. Ε, ο κύριος Αντόρ ήταν εδώ χθε, ο Επίτροπος, ε, και εγκρίθηκε από την Επιτροπή η απόφαση. Όσοι από εσά λοιπόν δεν έχουν διαβάσει την ανακοίνωση, Α γνωρίζουν ότι πρόκειται για ενσωματωμένες, ε, ολοκληρωμένε κατευθυντικές γραμμέ, Μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής και ε, έστειλα σήμερα στους κοιόδης εισηγητές ε, αντίγραφο του κειμένου και σημείωσα, διότι αυτό είναι επιβεβαίωση σε αυτά που έχω πει νωρίτερα, ότι θα ε, ε, έχω διαβουλεύσεις με τους ε, σκιώδεις προτού να υποβάλω προς μετάφραση το κείμενο. Εάν λοιπόν έχετε παρατηρήσει, εάν έχετε κάτι που θέλετε να συμπεριληφθεί στο κείμενο, υπάρχει η δυνατότητα. Κατόπιν θα συνεχίσουμε στις, με την εξέταση των τροπολογιών. Κάποιες παρατηρήσεις επιτρέψτε μου. Θα δείτε ότι η έκθεση είναι πολύ γενική, κάτι που οφείλεται στο γεγονό ότι οι κατευθυντήρε γραμμέ, στη μορφή που έχουν θέτουν στόχου κατευθύνσεις προ τι οποίε θα πρέπει να κινηθούν τα κράτη-μέλη. Ο τρόπο εφαρμογή θα πρέπει να καθοριστεί από τα ίδια τα κράτη-μέλη. Από την άλλη, το κείμενο προσπαθεί να αποφύγει οποιαδήποτε αναφορά στη χρηματοδότηση. Αυτό το αφήνουμε στα κράτη-μέλη και γίνονται κάποιε νήξει ε, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, αλλά ουσιαστικά μόνο μία πρόταση κάνει αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Φαίνεται λοιπόν ότι το κείμενο αποφεύγει ε, θέματα χρηματοδότηση που είναι πρόβλημα και αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε στην έκθεσή μα, διότι θέλουμε να υιοθετήσουμε τι ολοκληρωμένε κατευθυντήριε γραμμέ ω ε, μέρο τη στρατηγική του 2020 το Σεπτέμβριο. Πώ θα το κάνουμε αυτό όμω, εάν δεν γνωρίζουμε τίποτα σχετικά με τη χρηματοδότηση. Θα δεσμευτούμε. Πώ μπορούμε να δεσμευτούμε χωρί να ανοίξουμε συζήτηση σχετικά με το ε, χρηματοοικονομικό πλαίσιο, το δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, το πρόβλημα αυτό φαίνεται στο κείμενο, γι' αυτό είναι τόσο γενική η διατύπωσή του. Από την άλλη, το κείμενο περιέχει πολλές ε, περιτολογίες, ε, επαναλαμβάνει μέχρι 4-5 φορές τα ίδια πράγματα. Το προήμιο αναφέρεται σε όλα τα κεφάλαια, αλλά ε, στις κατευθυντήριες γραμμές βλέπουμε να επαναλαμβάνεται κατά λέξη το ίδιο κείμενο που έχει πάρθει από αλλού. Με copy-paste έχει γίνει όλη αυτή η δουλειά. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να χτενιστεί το κείμενο. Δεν υπάρχει λόγος να επαναλαμβάνουμε πράγματα. Άλλη παρατήρηση. Σημαντικά στοιχεία λείπουν από το κείμενο. Η πολιτική συνοχή, για παράδειγμα, θα πρέπει να τονιστεί και γίνεται αναφορά στην ε, περιφερειακή, οικονομική και κοινωνική συνοχή που υποτίθεται ότι είναι σημαντικό μέρος των κατευθυντήριων γραμμών. Αυτό είναι όμως το μόνο η μόνη, η μόνη σχετική αναφορά σε ένα κείμενο ανεπαρκέ. Α κοιτάξουμε τώρα τι ίδιε τι κατευθυντήρε γραμμέ. Η νέα στρατηγική Υπόθηκε ότι 24 κατευθυντήριες γραμμέ είναι υπερβολικά πολλέ. Θα πρέπει λοιπόν να, σκεφτούμε, ε, να συγκεντρωθούμε σε 10, από τις οποίες οι 4 θα έχουν να κάνουν με την απασχόληση. Υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την ορολογία, διότι λέμε ότι θα πρέπει να περιοριστεί, να μειωθεί η ε, ανεργία που οφείλεται σε δομικά προβλήματα, σε διαφορετικά προβλήματα. Δεύτερον, ε, λέμε ότι θα πρέπει να παρέχονται να παρέχει τη δυνατότητα απόκτηση ε, δεξιοτήτων που να είναι σχετικέ με την ε, αγορά εργασία, που να ενδιαφέρουν την αγορά εργασία ε, τη διαβίω εκμάθηση κτλ. Μιλάμε για τι κατευθύνσει γραμμέ 7, 8, 9. Λέμε ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα του εκπαιδευτικού συστήματο. Μιλάμε για τη διαβίω εκμάθηση. Ε, μου φαίνεται ότι οι δύο αυτέ κατευθύνσει γραμμέ αναφέρονται στο ίδιο θέμα. Δεν είναι σαφές γιατί έχει γίνει η επανάληψη αυτή. Η 10 δεν αφορά αποκλειστικά την απασχόληση. Μιλάμε για την καταπολέμηση τη στόχιας μιλάμε για την κοινωνική ένταξη. Δεν μπορεί να σημειωθεί πρόοδο στον τομέα αυτό χωρί τη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Υπάρχει λοιπόν λογικό σύνδεσμο. Διότι η καταπολέμηση τη φτώχεια ε, συνδέεται με τη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Κατά τα άλλα όμω φαίνεται να είναι ξένο στοιχείο στο σύνολο του κειμένου. Υπάρχει λοιπόν αρκετή δουλειά που πρέπει να γίνει πάνω στο κείμενο αυτό. Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να πω σε κάποιες λεπτομέρειε. Αναφερόμαστε σε 10 κατευθυντήριε γραμμέ. Οι ολοκληρωμένε κατευθυντήριε γραμμέ για τη στρατηγική 2020 θα αποτελέσουν τη βάση της στρατηγικής αυτής σύμφωνα με το κείμενο. Γι' αυτό θα πρέπει να εφαρμοστούν και να υιοθετηθούν μαζί με τη στρατηγική 2020. Στη χθεσινή συζήτηση συμφώνησα με την κυρία Μπερές ε, σε αυτά που είπε στον κύριο Αντόρ. Είναι αδύνατο να πετύχουμε τους στόχους ε, στην ε, Κομισιόν και στο Συμβούλιο. Αυτά αποφασίστηκαν χωρίς σεβασμό των δικαιωμάτων των ε, Ευρωβουλευτών, το να εργαστούν στη γλώσσα τους και να συμβουλευτούν τους δικούς τους εμπειρογνώμονες. Υπάρχει λοιπόν εδώ ένα θεμελιώδες πρόβλημα. Παρά το γεγονός ότι Μόλι τέλη Σεπτεμβρίου θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε θέση στο Κοινοβούλιο πάνω στι τις γραμμέ. Δεν μπορούμε να εργαστούμε πιο γρήγορα. Παρόλα αυτά, το Συμβούλιο θα υιοθετήσει πιο γρήγορα κάποιο κείμενο. Θέλουν λοιπόν να δημιουργήσουν ένα ανύπαρκτο καθεστώς. Επισήμως μιλάμε για κατευθυντήρες γραμμές που αποφθύνονται στα κράτη-μέλη, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να συνεχιστεί, διότι αυτό παραβιάζει τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου. Δεν επιτρέπεται η διαβούλευση ούτε με τους ενδιαφερομένους ούτε με τα εθνικά κοινοβούλια. Πρόκειται λοιπόν για ένα θεμελιώδες πρόβλημα. Ας εξετάσουμε λοιπόν τώρα τις κατευθυντήριες γραμμές. Σταθερότητα του οικονομικού συστήματος. Θέλουμε να εξαλείψουμε τις ανισορροπίες στην μακροοικονομία για να καταπολεμήσουμε προβλήματα ανισορροπίας εντός της Ευρωζώνης. Έχουμε τον τομέα της έρευνας της ανάπτυξης, ε, μας ενδιαφέρει η απόκτηση δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων. Μιλάμε για την ψηφιακή κοινωνία στο σημείο 4. Θέλουμε πιο αποτελεσματική ανάπτυξη. Ε, θέλουμε να εξετάσουμε, θέλουμε βιώσιμους πόρους, πράσινη η οικονομία, θέλουμε ε, μείωση των εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακα, όπως αναφέρει η κατευθύντα γραμμή 6 και θέλουμε να εξυγχρονίσουμε την βιομηχανική βάση. Όλα αυτά καλά. Η κατευθυντήρια γραμμή υπαριθμών 7 είναι η πρώτη κατευθυντήρια γραμμή που αναφέρεται στην απασχόληση. Ε, πρέπει να αυξηθεί η απασχόληση. Η 8 αναφέρεται στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης υψηλής ποιότητας ε, που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ε, αγοράς εργασίας. Αναφερόμαστε στη διαβίω εκμάθηση στην ε, απόκτηση δεξιοτήτων για θέσεις απασχόλησης υψηλή ποιότητα. Η κατευθυντήρια γραμμή 9 αναφέρεται στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην επαγγελματική κατάρτιση. Θέλουμε να αυξήσουμε την ποιότητα της εκπαίδευσης, να αυξήσουμε τη συμμετοχή και η 10 αναφέρεται στην καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης. Σαν μάντρα επαναλαμβάνονται τα ίδια πράγματα στο κείμενο. Το κείμενο μιλάει για έξυπνη, βιώσιμη, ενταξιακή ανάπτυξη, αλλιώς δεν μπορούν να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης. Ε, το κείμενο λέει ότι χρειάζονται φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις, ε, αναφέρεται στη διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας και, την, και της βιωσιμότητας των οικονομικών συστημάτων. Αυτά αναφέρονται και στις κατευθυντήρες γραμμές για την απασχόληση η υπό την ίδια μορφή. Αν γυρίσετε σελίδα βλέπετε ότι μιλάμε για εκπαίδευση, κατάρτιση ποιότητας και σε παρένθεση γίνεται αναφορά στη συνοχή, χωρίς όμως να γίνονται συγκεκριμένες αναφορές. Τα κράτη-μέλη καλούνται να εφαρμόσουν τις μεταρρυθμίσεις. εάν θέλετε να πούμε σε λεπτομέρειες, να πω ότι δεν μπορούμε να προοδεύσουμε έτσι. Το σημείο 7 που αναφέρεται στην αύξηση της συμμετοχής στην ε, αγορά εργασίας και στη μείωση της ε, ανεργίας που οφείλεται σε δομικά προβλήματα, ε, αναφερόμαστε και στην ελαστασφάλεια, το flexicurity. Λέμε ότι θα πρέπει να βασιστούμε στα συστήματα των μελών, θα πρέπει να μειωθεί η ανεργία που οφείλεται σε δομικά προβλήματα και θα πρέπει ε, γίνεται αναφορά στα ευέλικτε στις ευέλικτες συμβάσεις εργασίας, στη διαβιακμάθηση ε, και στην ε, μεταρρύθμιση των προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας. Πράγμα που δεν σημαίνει η επέκτασή τους. Μιλάμε για οικονομική σταθερότητα. Θα πρέπει οικονομική και η κοινωνική σταθερότητα να παρέχεται σε όλους. Ενώ η όλη λογική του συστήματος είναι μία προσέγγιση που βασίζεται στις οδηγίες. Δεν έχουμε υπότομα από κάτω προς τα πάνω, από τη βάση προς τα πάνω. Όσον αφορά την ευελιξία, Έχουμε εδώ μια πιο αναλυτική προσέγγιση. Μιλάμε για ε, συμβάσεις ε, μη χαρακτηριστικές. Ε, αναφερόμαστε στους αυτοαπασχολούμενους και θα πρέπει να δημιουργηθούν νέοι κανόνες για τις συγκεκριμένες αυτές ομάδες. Πιστεύω ότι αυτός ο στόχος είναι πολύ καλός. Κάποιες κοινωνικές ομάδες αναφέρονται, οι οποίες θα πρέπει να βοηθηθούν όσον αφορά την πρόσβασή του στην αγορά εργασία, όπω είναι οι νέοι, οι ηλικιωμένοι, οι άνθρωποι με αναπηρίε. Και όλοι όσοι έχουν ξεφύγει από την αγορά εργασίας. θα πρέπει να βελτιωθούν κάποια μέρη, ε, όπως και τα κείμενα που αναφέρονται στην, το σημείο του κειμένου που αναφέρονται στην ψηφιακή κοινωνία. Έχουμε εδώ και μια καινοτομία. Καλούνται τα κράτη-μέλη να αναθεωρήσουν τα οικονομικά τους συστήματα και τα φορολογικά τους καθεστώτα. Αυτό είναι μια αναφορά στα φορολογικά προγράμματα των κρατών μελών τι βάρη θα πρέπει να φέρουν οι εργαζόμενοι στην αγορά εργασίας και πώς μπορούμε να τους ανακουφίσουμε από τα φορολογικά βάρη. Από την άλλη αναφέρεται και η ισότητα ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες. Θα πρέπει η ίδια εργασία να μείβεται με τον ίδιο τρόπο. Επίσης αναφερόμαστε στους νέους, τα άτομα με αναπηρίες και τους νόμιμους μετανάστες. Αυτοί αναφέρονται στο κείμενο. Χθες είχαμε συζήτηση για το συγκεκριμένο αυτό θέμα. Έχουμε και τους αυτοαπασχολούμενους. Έχουμε κάποια νούμερα, κάποια στοιχεία στον τομέα αυτών. Για την ηλικιακή ομάδα 20 με 64 ετών, ε, ο στόχος της Λισαβόνας ήταν ε, το 70% για την απασχόληση, τώρα πια είναι 75% και για τους άντρες και για τις γυναίκες, όπως προτείνεται στο κείμενο της Κομισιόν. Αυτό επαναλαμβάνεται και στη στρατηγική 2020. Στα 17 χρόνια δηλαδή θα πρέπει να πετύχουμε απασχόληση ύψους 75% στην Ευρώπη. Η επόμενη κατευθυντήρια γραμμή έχει να κάνει με την παραγωγικότητα και την αύξηση της απασχολησιμότητας, την πρόθεση νέων δεξιοτήτων, την εκπαίδευση και την διαβίου εκμάθηση. Με άλλα λόγια θα πρέπει ο καθένας να λαμβάνει μια δεύτερη ευκαιρία προσχώρησης ένταξης ε, στην ε, αγορά εργασίας. Θα πρέπει να υπάρχει αναγνώριση κάποιων δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων. Θα πρέπει επίσης να εξαλειφθούν τα εμπόδια στην κινητικότητα. Θα πρέπει λοιπόν να εξαλειφθούν τα εμπόδια. Είναι εξαιρετική ιδέα αυτή δεν ε, ε, ε, διευκρινίζεται αναλυτικά όμως στο κείμενο. Ουσιαστικά μιλάμε για προώθηση των ανθρώπων χωρίς προσόντα, των ηλικιωμένων, των νέων. Δεν θέλω να επαναλάβω όλα όσα αναφέρονται στο κείμενο. Η κατευθυντήρια γραμμή επίσης αναφέρεται στην εκπαίδευση. Δεν έχω καταλάβει, ε, δεν έχω καταλάβει γιατί επαναλαμβάνονται αυτά τα πράγματα στο κείμενο. Αναφερόμαστε στα εκπαιδευτικά συστήματα, σε όλα τα, σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος, τα οποία θα πρέπει να προωθηθούν. Θα πρέπει να βελτιωθεί η συμμετοχή στην ανώτατη εκπαίδευση. Αυτό είναι γνωστό σημείο της στρατηγικής 2020. Επαναλαμβάνονται λοιπόν τα ίδια στοιχεία και οι ίδιοι στόχοι. Θα πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των ανθρώπων που εγκαταλείπουν το σχολείο νωρίτερα. Κάθε επίπεδο του εκπαιδευτικού συστήματος θα πρέπει να παρέχει ε, προσόντα και δεξιότητες ε, που να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. η συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να αυξηθεί από 10% σε 40%. Λίγα λόγια τέλος. Για την τελευταία κατευθυντήρια γραμμή, που αναφέρεται σε μια κοινωνία ένταξης και στη καταπολέμηση της στόχιας. Ανακύπτουν εδώ οι γνωστές ιδέες. Θέλουμε σημαντική μείωση της φτώχειας. Το κείμενο αυτό δεν αναφέρει δείκτες που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κανείς για να μετρήσει την επιτυχία των στόχων. Τον να αναφερόμαστε στην καταπολέμηση των διακρίσεων, στην κατευθυντήρια αυτή γραμμή. Πάλι το κείμενο αναφέρει την διαβίω εκμάθηση. και αναφέρει ότι όλοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Τα καθεστώτα και συστήματα κοινωνικής πρόνοιας θα πρέπει να αναθεωρηθούν και θα πρέπει να διασφαλίζεται η οικονομική ισορροπία εντός των συστημάτων αυτών. Αναφέρονται και οι ομάδες στόχοι στις κατευθυντήριες γραμμές αυτές. Οι πιο φτωχοί φαίνεται να κινδυνεύουν περισσότερο από, από τον κοινωνικό αποκλεισμό. Μιλάμε για μονογονεακές οικογένειες, για άτομα με ειδικέ ανάγκες, νέους, παιδιά, ηλικιωμένους, νόμιμους μετανάστες και άτομα με αναπηρίες. Και πάλι έχει θεθεί μειωθεί ο αριθμός των φτωχών κατά 25% δηλαδή κατά 20, συγγνώμη, κατά 20 εκατομμύρια άτομα σύμφωνα με το κείμενο. Το κείμενο αυτό λοιπόν είναι πολύ γενικό, έχει πολλές περιτολογίες, επαναλαμβάνεται συνεχώς και δεν εξηγεί αναλυτικά τα πράγματα, πράγμα κατανοητό διότι είναι άγνωστες αυτή τη στιγμή οι δημοσιονομικές προϋποθέσεις. Έχω επίσης την εντύπωση ότι δεν γίνεται αρκετή αναφορά στην πολιτική συνοχής. Μη σας μιλήσω για νούμερα και στοιχεία, δείκτες που βοηθούν στη μέτρηση της απόδοσης. Δεν αναφέρεται η πολιτιστική πολιτική ούτε το σημαντικό θέμα της απασχολησιμότητας. Είναι σημαντικός παράγοντας και η κοινή γεωργική πολιτική είναι σημαντικό μέσο στα χέρια της κοινότητας για την αύξηση της απασχολησιμότητας και την οικονομική ανάπτυξη. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο υποβολής τροπολογιών και ε, βελτιώσεων για το κείμενο. Σας ε, παρακαλώ λοιπόν να εξτάσετε το κείμενο, το οποίο από σήμερα θα είναι διαθέσιμο. Την Τρίτη θα υποβάλω το δικό μου κείμενο για μετάφραση. Μέχρι τότε είμαι ανοιχτός, είμαι διαθέσιμος για να έχω διαβουλεύσεις με τους κοιόδης εισηγητές και όσους από εσά Ε, θέλουν. Ε, όσοι δεν έχετε, ε, δεν έχετε συμβάλει μέχρι τότε θα έχετε τη δυνατότητα αργότερα να συμβάλλετε στο κείμενο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τούρινεν. Ωραία. Ωραία, δουλεύει τώρα το μικρόφωνο. Ευχαριστώ κύριε Όρη και επίσης την κυρία Μπερές που όρθωσε το ανάστημα του Κοινοβουλίου εκ μέρου μα όσον αφορά τι κατευθυντήριε γραμμέ. Θα πρέπει να πούμε ότι όντως μας παρέκαμψαν σε αυτήν εδώ την υπόθεση και σας ευχαριστώ που μπορέσατε να σταθείτε ε, ε, και στο ύψος των περιστάσεων για την υπόλοιπη διαδικασία. Εγώ αναρωτιέμαι ποια είναι η λογική που κρύβεται πίσω από τις αλλαγές που είδαμε σε σχέση με τις πρώτες κατευθυντήριες και τις τωρινές. Όπως είπε ο κύριος Έρη, υπάρχουν πολλά λόγια, αλλά πολύ λίγες λεπτομέρειες, συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά ξέρω ότι η συνάδελφος θα αναφέρει περισσότερα. Αυτό που ήθελα να πω και που με κάνει να συμφωνώ με τον κύριο Όρη που το ανέφερε, είναι ότι θα πρέπει να συνδεθεί με τον προϋπολογισμό και τη χρηματοδότηση. Αυτό θα ήταν ένα πολύ σημαντικό σημείο για μας. Επίσης, θα θέλαμε να έχουμε πιο συγκεκριμένους στόχους και μέτρα για την νεότητα, για τον κοινωνικό αποκλεισμό που αναφέρεται λίγο. Ξέρω την έντονη διατύπωση, αλλά πραγματικά πιστεύω πως χρειάζεται να γίνει μια ε, τίμια συζήτηση επ' αυτού. Στις δυτικές χώρες έχουμε ε, μείωση των ε, μισθών, έχουμε πτώση των προδιαγραφών ε, στον τομέα της υγείας, έχουμε αύξηση της μαύρης αγοράς εργασίας. Αυτό δεν είναι κοινωνική Ευρώπη. Θα πρέπει να το καταπολεμήσουμε τόσο μέσω των νομοθεσιών μας, όσο και μέσω της επιβολής των όσων αποφασίζουμε. Δηλαδή θα χρειαζόταν μια πραγματική ατζέντα για αξιοπρεπή δουλειά και επίση γιατί ε, την φτώχεια δεν μπορούμε να την καταπολεμήσουμε μόνο μέσω της απασχόλησης. Ξέρουμε πως υπάρχουν 18 εκατομμύρια εργαζόμενοι φτωχοί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Δηλαδή απασχόληση δεν είναι η μόνη απάντηση. Πιστεύω επίσης πως θα πρέπει να υπάρχει ισχυρότερη σύνδεση ανάμεσα στις ε, κατευθυντήριες για την απασχόληση και τις κατευθυντήριες για την οικονομία λέει πολλά για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση, αλλά δεν λέει τίποτα για το πώς θα γίνουν όλα αυτά και πώς θα πρέπει να δεσμευτούν για αυτή τη διαδικασία. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε πολύ ισχυρή πολιτική επενδύσεων. Πολύ δουλειά λοιπόν υπάρχει ακόμα να γίνει, πρέπει ακόμα να γίνει και συμφωνώ με τον κύριο Όρη και τον ευχαριστώ γιατί έχει ανοιχτό μυαλό και ελπίζω πως η διαδικασία θα είναι θετική γιατί η Επιτροπή μας μπορεί να προσθέσει στοιχεία ποιοτικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα. Σε 10 λεπτά πρέπει να έχουμε τελειώσει τη συζήτηση. Θα έχετε την ευκαιρία από τη στιγμή που θα έχει ε, συντάξει την εκθεσία του φαντάζομαι στις 17 Μαΐου να, να μπείτε σε περισσότερες λεπτομέρειες όταν θα δείτε το γραπτό κείμενο. Για την ώρα έχω 5 ακόμα μιλητέ, ε, οπότε παρακαλώ να είστε όσο γίνεται πιο σύντομοι για να ολοκληρώσουμε την ατζέντα μας ε, χωρίς να αφήσουμε τίποτα. Η κυρία Κορνέλησεν. Σας ευχαριστώ. Εγώ νομίζω πως ε, όλες αυτές οι προτάσεις ε, χρησιμοποιούν απλά κάποιες νέες καραυγαλές λέξεις χωρίς όμως ε, συγκεκριμένα μέτρα. Μια καλή συγκεκριμένη πολιτική σημαίνει στόχους, χρήματα και κυρώσεις. Και επίση, ε, εδώ βλέπουμε ας πούμε, το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση, για το Κοινωνικό Ταμείο που σχετίζονται με την απασχόληση, αλλά θα έπρεπε στο πλαίσιο της Ευρώπης 2020 θα έπρεπε να εξετάσουμε όλες τις ευρωπαϊκέ δαπάνε και να τις ανακατευθύνουμε προς την ίδια τον ίδιο προορισμό ώστε να έχουμε αποτελέσματα. Για να πετύχουμε αποτελέσματα θα πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι τα αποτελέσματα. Πραγματικά θα έπρεπε να έχουμε καλούς και διαφοροποιημένους στόχους, καθώς και τους σωστούς χρήστες που θα μας ε, δείξουν αν επιτύχαμε τους στόχους αυτούς. Ένα παράδειγμα, οι κάτω χώρες στη στρατηγική της Λισαβόνας έθεσαν το στόχο ε, για την απασχόληση των γυναικών. Τα κατάφεραν πολύ καλά να πετύχουν το στόχο, αλλά μέτρησαν ακόμα και τις γυναίκες που δουλεύουν ένα δύο την ημέρα. Αυτό δεν έχει να κάνει με πλήρη απασχόληση ή για ε, δεν είναι σωστό για την καταμέτρηση και τη στόχη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ που ήσασταν σύντομοι. Η κυρία Γκόντς. Σας ευχαριστώ. Θα είμαι και εγώ σύντομη. Το κείμενο αυτό είναι όντως πολύ γενικόλογο. Δεν μπορεί κανείς να καταλάβει πώς θα προχωρήσει η εφαρμογή. Το βασικό πρόβλημα, νομίζω, έγκυται στο γεγονό ότι οι οικονομικές κατευθυντήριες γραμμές, οι κατευθυντήριες γραμμές απασχόλησης και, και οι κατευθυντήριες για τη φτώχεια δεν είναι αρκετά ολοκληρωμένες. Θέλουμε να βελτιώσουμε την απασχόληση, αλλά χωριστά μιλάμε για την κατάρριξη των διακρίσεων, ενώ το ένα συνδέεται στενά με το άλλο. Μιλάμε για τη βελτίωση της ποιότητας της ε, παιδείας και μετά Χωριστά μιλάμε για την παιδική φτώχεια και τη δύσκολη κατάσταση των οικογενειών, ενώ τα δύο αυτά συνδέονται στενά. Θα πρέπει η παιδεία να ξεκινά σε ένα πολύ ε, πρώιμο στάδιο, γιατί οι δεξιότητες καθιστούν τους νέους πιο ικανούς για την ε, αγορά εργασίας. Έπειτα, δεν υπάρχει τρόπος μέτρησης. Μιλάμε για διακρίσεις για την πολιτική συνοχή, η πολιτική συνοχή και ανανέωσή της είναι κλειδί, θέμα κλειδί για να τα καταφέρουμε και είναι πολύ δύσκολο να δούμε πώς όλα αυτά συνδέονται. Τώρα, το... η κατευθύντρια 7 Μια επισφαλή εργασία είναι επίση πρόβλημα, αλλά δεν έχω και χρόνο για να σα τα αναλύσω όλα, θα τα ξανασυζητήσουμε ευτυχώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ελέγχθησαν ήδη κάποια πράγματα. Υπάρχουν ορισμένε θετικέ προσεγγίσει στι κατευθυντήριε αυτέ γραμμέ, αλλά κατά τα άλλα είναι πολύ θολέ και ανακριβεί. Και έλπιζα ότι πραγματικά θα ήταν εξαιρετικέ, γιατί χρειάστηκε μεγάλο χρονικό διάστημα για να εκπονηθούν. Ε, θεωρώ ότι απουσιάζει εδώ ο στόχος της πλήρους απασχόλησης. Πρέπει να διατυπωθεί ρητά, γιατί δεν έχουμε εδώ καθόλου φιλόδοξους στόχους. Και αυτό σημαίνει ότι παραγωνίζουμε πάρα πολλούς ανθρώπους, αφήνουμε στην άκρη. Αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή τελικά στοχεί στην εκπλήρωση της πολιτικής της. Ο Επίτροπος χθε είπε ότι θέλει να μειώσει την ανεργία, αλλά δεν μας είπε πώς προτίθεται να το κάνει. Και εγώ συμμερίζομαι την άποψη ότι θα πρέπει να μεριμνήσουμε ότι θα υπάρξουν ε, ποιοτικέ θέσει εργασία. Δεν θέλουμε πλήρη απασχόληση πάση θυσία, όχι με εκμετάλλευση ε, εργαζόμενων με χαμηλέ αποδοχέ, επισφαλεί θέσει εργασία κλπ. Προσωρινή απασχόληση κλπ. Ε, θα πρέπει να κατορχυρώσουμε την πλήρη απασχόληση με ένα σωστό τρόπο. Θα πρέπει, και αυτό ήδη υπόθηκε από τους συναδέλφους, να εξασφαλίσουμε επενδύσει για την κατοχήρωση μόνιμων θέσεων εργασίας και για τη δημιουργία νέων θέσεων. Θα πρέπει να λάβουμε να, εξετάσουμε μέσα που να μας βοηθήσουμε να εξέλθουμε από την κρίση. Για παράδειγμα, η πολιτική της συνοχής. Η κατευθύνια γραμμή υπαριθμών 7 ξεκινά αυτής εξ αρχής με το Flex Security. Ε, θεωρώ ότι είναι άστοχο σε μια τέτοια τύπωση πολιτικής απασχόλησης να ξεκινάει κανείς με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι ε, στην κρίση έχουν γίνει αντικείμενο εκμετάλλευση οι εργαζόμενοι και ο Επίτροπος αναφέρθηκε σε αυτές τις ε, προποθέσει προποθέσει σε ολόκληρη την Ευρώπη και είπε ότι θα πρέπει να προσεγγίσουμε το θέμα αυτό. Στη Γερμανία τα πράγματα είναι τόσο διαφορετικά όταν μιλάει για την flexicurity από τις άλλες χώρες. Όσον αφορά τη μείωση της διαθετικής ανεργίας, εδώ θα πρέπει να γίνουμε, γίνουμε πολύ πιο συγκεκριμένοι και να δούμε τα πράγματα πολύ πιο διαφοροποιημένα, περισσότερες αποχρώσεις. Το είπαν οι συνάδελφοι, χρειαζόμαστε χρόνο να πούμε σε ποιο τομέα θέλουμε να παρέμβουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Για παράδειγμα, οι νέοι ο κύριος Μαν χθε είπε ότι θα ήταν άδικη παρέμβαση στην πολιτική των χωρών μελών. Αλλά εγώ πιστεύω ότι η Επιτροπή στοχεύει μόνο στον ανταγωνισμό. Αλλά ο ανταγωνισμός ταιριάζει ακριβώς, ενδείκνεται εδώ στην εκπλήρωση αυτών ακριβώς των στόχων. Τέλος, όσον αφορά την εξειδίκευση. Ναι, η εξειδίκευση είναι σημαντική. Γιατί... Ε, θέλουμε μόνο αυτό το, την αυτού του στόχου. Ξέρουμε ότι υπάρχουν 10% ε, των μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο. Η κατευθύρια γραμμή 10 αναφέρθηκε επίσης για την καταπολέμηση της φτώχειας. Σημαντικό είναι η καταπολέμηση της φτώχειας των ίδιων των εργαζόμενων. Επίσης θα πρέπει να κλείσουμε κάποια χάσματα στι θέσει εργασία, Για παράδειγμα, όταν στη Γερμανία ε, οι εργαζόμενοι πληρών, οι εργοδότες πληρώνουν μέσω των κρατικών επιδοτήσεων, χρηματοδοτούν μέσω των κρατικών επιδοτήσεων τις θέσεις εργασίας. Με αυτό συνέδεται το θέμα της μεταρρύθμισης των κοινωνικών συστημάτων και από την άλλη το αίτημα για την ε, σταθεροποίηση του προπολογισμού στο επίπεδο των χωρών μελών. Ε, Όλα αυτά είναι δύσκολα, αλλά νομίζω ότι η κοινωνική ισορροπία στην Ευρώπη θα πρέπει να εδρεωθεί. Δεν είναι εδώ να συνεχίσουμε στο πλοίο αυτή τη ανισορροπία. Θα πρέπει να αλλάξουν κάποια βασικά πράγματα στι κατευθυντήριε γραμμέ. Ε, μετά από όλα όσα ακούσαμε από του συναδέλφου μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα πετύχουμε αυτέ τι βελτιώσει. Έχουμε δύο ακόμα μιλητές αλλά ήδη δυστυχώ έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μα. Κυρία Χάρκιν, θα είμαι πολύ σύντομη. Ε, σύμφωνα με τον κύριο Ρή, ε, έδωσα μια, έκανα μια βιαστική, έδωσα μια βιαστική ματιά στι κατευθυντήρε γραμμέ η έννοια κατάρτιση εμφανίζεται οκτώ φορές. Ε, υπάρχουν πάρα πολλές επικαλύψεις εδώ. Συμφωνώ με τους στόχους που, θέθη, που τέθηκαν, αλλά το ερώτημά μου και εμένα είναι το πώς μπορούν να γίνουν όλα αυτά. Χρειαζόμαστε μια εντονότερη διασύνδεση μεταξύ απασχόλησης και οικονομικών κατευθυντήριων γραμμών. Για παράδειγμα, η γραμμή 4 που μιλάει για την καινοτομία ε, και για, την, ε, για το δημοτικό της ψηφιακής οικονομίας. Όλα αυτά συνδέονται με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και νομίζω το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε καλύτερες ευκαιρίες για τους επιχειρηματίες. Θα πρέπει να υπάρξει μια στενότητα διασύνδεση μεταξύ όλων αυτών των πτυχών. Ε, ε Νομίζω ότι όλα αυτά είναι κάπω αόριστα. Δεν είναι αρκετά συγκεκριμένα, δεν συνδέονται με τον προπολογισμό. Για παράδειγμα, το κοινωνικό ταμείο που είναι από τα σημαντικά εργαλεία που έχουμε αναφέρεται μόνο μία φορά δεν ε, βλέπω πουθενά να αναφέρεται το τομείο παγκοσμιοποίηση η συνοχής. Ε, ε, συμφωνώ με του προηγούμενου ομιλητέ, Χρειάζεται να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στου νέους και στου ε, εργαζόμενους που δεν έχουν επαρκή αποδοχή. Νομίζω ότι είναι αρκετά ισχνές οι κατευθυντήρες αυτές γραμμές. Ο κύριος Χάντλ. Ε, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, θεωρώ ότι έχουν δίκιο οι προλαλήσινε και ίσω είναι μέλημα της δικής μας πολιτική ομάδα να είμαστε λίγο πιο τολμηροί στη διατύπωση. Θα ήθελα να το πω ξεκάθαρα. Ε, ε με αυτό το έγγραφο μπορεί ο καθένας ε, να κάνει ό,τι του περνάει από το κεφάλι και από την άλλη δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Εάν ισχύει ότι η Eurostat το ευρωπαϊκό δυναμικό απασχόλησης κατά 60% τοποθετεί σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας και πολλοί θεωρούν ότι η κοινωνική συνοχή στις χώρες μέλη ε, απειλείται εξαιρετικά από αυτές τις τάσεις και τις εξελίξεις, θα πρέπει νομίζω η Επιτροπή να βρει μια απάντηση μέσω αυτών των κατευθυντήριων γραμμών. Και δυστυχώ δεν γίνεται μέσω αυτού του εγγράφου. Δεύτερον, όταν μιλάμε για τη flexicurity με ένα κριτικό τρόπο σε ολόκληρη την Ευρώπη, γιατί έχουμε πάρα πολύ ευελιξία αλλά ελάχιστη ασφάλεια, νομίζω ότι δεν ε, είναι αρκετή μια φράση σε σχέση με το πρόβλημα αυτό που αναφέρεται στο έγγραφο αυτό. Τώρα όσον αφορά τι αποφάσει του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, εδώ υπονομεύεται ο κοινωνικό διάλογο γιατί υπονομεύονται θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων. Νομίζω ότι οι κατευθυντήριε γραμμές θα πρέπει να είναι πιο ξεκάθαρες για το μέλλον όσον αφορά με το δικαίωμα συναπόφαση που θα πρέπει να συνοδεύουν τον κοινωνικό διάλογο. Και τέλος, τι γίνεται με μια πολιτική η οποία θεωρεί την κοινωνική πρόοδο στην Ευρώπη υπό τη μορφή ενός ε, ανταγωνισμού και τελικά το συρεκνώνει σε μια ε, κοινωνική ε, ρήτρα. Αυτά είναι τρία σημεία τα οποία απουσιάζουν εδώ και ως ε, σκιώδης εισηγητές θα έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε με την επεξεργασία αυτού του κειμένου. Ο Τόμας Μαν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ναι, ε, τα όσα είπε ο προηγούμενος ομιλητής ίσως έχει δίκιο όταν αναφέρθηκε σε κάποιους ε, ιερωμένους και θεωρητικούς Νομίζω ότι η Ρώμη σε πολλά πράγματα πήγε πολύ μακρύτερα από ό,τι αποτολμούν ε, να το πράξουν ορισμένε χώρες ε, μέλη. Ε, ο συνάδελφος Στάινμπρουκ επεσήμενε ότι χθε είχα μια διαφορετική άποψη από εσά. Νομίζω δεν υπάρχει τόσο μεγάλη απόκληση. Εγώ απλώ ε, έθεσα στον Επίτροπο το ερώτημα ποιε είναι οι ευκαιρίε υλοποίηση αυτού του προγράμματο εκ μέρου τη Επιτροπή ώψη του γεγονότο ότι οι χώρε ε, μέλη τελικά φοβούνται το θέμα της ε, ποσοτικοποίηση ή τη αναφορά τη δήλωση κάποιων αριθμών. Αυτό το θέμα έθεσα. Νομίζω ότι είναι καλύτερο να υπάρξει στενότερη συνεργασία. Νομίζω ότι δεν είναι καλό να θέσουμε αυτούς τους υποψηφίους σε ένα μαύρο ή κόκκινο κατάλογο, αλλά να πούμε ότι οι χώρες που, ήταν, ή που είχαν καλές επιδόσεις τελικά να επιβραβευθούν με έναν τρόπο. Νομίζω ότι αυτή είναι μια δυνατότητα και ίσως σε αυτό το σημείο δεν είμαστε δεν αποκλίνουμε τόσο πολύ. Τώρα, όσον αφορά το θέμα flexicurity, η συνάδελφο ε, Γκρινή έχει επεξεργαστεί το θέμα αυτό σε σχέση ακριβώ με τι άτυπε συμβάσει εργασία. Και βεβαίω όλα αυτά είναι αλληλένδετα και σχετίζονται και με τι κατευθυντήριε γραμμέ. Αλλά νομίζω ότι εδώ έχουμε τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε το θέμα τη ε, flexicurity. Και θα ήθελα να επισέλθω στο ζήτημα αυτό σε σχέση ακριβώ με αυτή την έκθεση. Τώρα, όσον αφορά το Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχή, ε, ήθελα να θέσω το ερώτημα στον Επίτροπο, αλλά δεν είχα τον αρκετό χρόνο. Ε, εγώ ρώτησα πώς είναι να υπάρξουν περισσότερα κονδύλια, γιατί τα κονδύλια, σε αντίθεση με άλλα κονδύλια που αποφασίζουμε στην Ευρώπη, είναι χρήματα τα οποία τελικά φτάνουν στον παραλήπτη στην Ευρώπη. Θεωρώ ότι το μοντέλο του Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου Συνοχής ήταν πετυχημένο. Και, ε, νομίζω ότι θα πρέπει να αποτελέσει μοντέλο για τις υπόλοιπες πολιτικές. Αυτά είπα στον ε, Επίτροπο και νομίζω ότι αν το πράξουμε μπορούμε όλοι να συνεργαστούμε και οι ομιλητές που προηγουμένως έβαλα, έλαβαν το λόγο. Η κυρία Κέπχαρτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Δεν έχω πολλά να πω. Σημείωσα προσεκτικά όλες τις παρατηρήσεις και προσλέπω στις προτάσεις των συναδέλφων. Θα προσπαθήσω να υποβάλω κείμενο που θα υποβάλω στους μεταφραστές το οποίο θα αποτελεί σημαντική βελτίωση σε σχέση με το κείμενο που έχουμε μπροστά μα. Ό,τι δεν μπορούμε να βελτιώσουμε αυτή τη στιγμή, μπορούμε πάντα να το κάνουμε αργότερα με την υποβολή τροπολογιών. Είτε μα αρέσει είτε όχι. Το θέμα αυτό είναι από τα πιο επίκαιρα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Θέλουμε λοιπόν καλύτερες, πιο χρήσιμες κατευθυντήρες γραμμές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ωρή. Πρωτού προχωρήσουμε στην επόμενη έκθεση θα ήθελα να καλωσορίσουμε μια ομάδα προσκεκλημένων ε, από το ΟΠΕΒΕΔΕΡ. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε. Το επόμενο θέμα μας είναι οι άτυπες συμβάσεις, εξασφαλισμένη επαγγελματική πορεία, ευελιξία με ασφάλεια και νέες μορφές κοινωνικού διαλόγου. Η κυρία Γκρίνη, παρακαλώ. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά αυτή την έκθεση πρωτοβουλία, θα ήθελα καταρχήν να σα επενθυμίσω ότι ο κανένα ε, παραμένει ε, η σύμβαση όλη τη ε, διάρκεια. Ωστόσο, θα πρέπει να μπορούμε να προσαρμοστούμε ε, στις νέες συνθήκες εργασίας και βεβαίως να διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν διάφορες μορφές σύμβασης στις διάφορες χώρες μέλη. Και νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια απάντηση πλαισιώνοντας αυτές τις συμβάσεις για να προλάβουμε τις καταχρήσεις τις οποίες αναφερθήκαμε. Και ε, φυσικά σε αυτές τις ε, τυπικές ε, συμβάσεις, χαρακτηριστικές συμβάσεις, θα πρέπει επίσης να διατηρήσουμε εκ την ευελιξία για τις επιχειρήσεις, αλλά επίσης και μια παροχή ασφάλειας στους εργαζόμενους οι οποίοι αποδέχονται αυτές τις συμβάσεις. Λοιπόν, στις τυπικές συμβάσεις θα πρέπει να συγκεντρώσουμε τις διάφορες μορφές εδώ να τις συνενώσουμε και νομίζω ότι η Επιτροπή μπορεί να μας προτείνει κάποιους τρόπους για να πλουστεύσουμε οτιδήποτε υπάρχει σήμερα και να λάβουμε επίσης κάποια παραδείγματα στο επίπεδο των διαφόρων χωρών μελών όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές. Νομίζω ότι θα πρέπει να στηριχτούμε εδώ και όσον αφορά τη Security, ε, συχνά αναφέρουμε τη Δανία, αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες που έχουν μορφέ συμβάσεων που θα μπορούσαν να είναι ενδιαφέρουσε για μα. Η κρίση επίση ε, προσέθεσε κάποια στοιχεία σε αυτή την ε, ζήτηση Security, δηλαδή άτυπων συμβάσεων. Έστω και αν σα υπενθύμισα τη βασική σύμβαση της αόριστης διάρκεια τη βασική συνθήκη συγγνώμη, της αόριστης διάρκειας για τις συμβάσεις. Αυτή είναι η θεμελιώδη συνθήκη ε, που ισχύει για τις συμβάσεις, θα πρέπει να ισχύει για τις συμβάσεις. Αυτό το οποίο διαπιστώνουμε στη Γαλλία είναι ότι όσο, πολύ, όσο περισσότερο μεγαλώνει ο, ο φόβος της ανεργίας, ε, τόσο περισσότερο ε, απαντώνται οι άτυπες μορφές σύμβασης που ε, λειτουργούν για κάποιο χρονικό, που ισχύει για κάποιο χρονικό διάστημα, για να μπορέσει κανείς να επανέλθει πιο γρήγορα στην αγορά εργασία. Τώρα, όσον αφορά την παράνομη εργασία, ίσω, εάν πλαισιώσουμε καλύτερα τι τυπικέ συμβάσει και να προτείνουμε διαφορετικών τύπων συμβάσεων, αυτό θα μα επιτρέψει ενδεχομένω να αποφύγουμε αυτές τις ε, μορφές παράνομη εργασία. Στο ζήτημα τη. flexicurity, ευελιξία για τις επιχειρήσεις όπως είπαμε, αλλά κυρίως ασφάλεια για τους ε, μισθωτούς. Και νομίζω ότι αυτό το στόχο εξυπηρετεί αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας. Φυσικά κατανοούμε ότι οι επιχειρήσεις και συγκεκριμένα ε, σήμερα ακόμα περισσότερο δυσκολεύονται να ε, στοχεύσουν μακροπρόθεσμα στην αγορά εργασίας και ε, δυσκολεύονται να προτείνονται συμβάσεις ε, αόριστης διάρκειας. Νομίζω λοιπόν ότι αυτές οι άτυπες συμβάσεις στο πλαίσιο της flexicurity πράγματι μπορούν να αποτελέσουν μια απάντηση ε, σε αυτή την κάπως δυσχερή περίοδο κρίσης, αλλά βεβαίως θα πρέπει να έχουν μεταβατικό χαρακτήρα. Τώρα, όσον αφορά την εξασφάλιση μιας επαγγελματικής σταδιοδρομίας, βεβαίως θα πρέπει να καταγγείλουμε την αντικατάσταση, την καταχρηστική αντικατάσταση των μόνιμων εργαζόμενων από άτυπα εργαζόμενους. Οι άτυπες αυτές συμβάσει βεβαίω μπορούν να επιτρέψουν σε ανθρώπους που δεν μπορούσαν να εργαστούν γιατί έχουν ε, διαφορετικές ανάγκες ίσως θα μπορούσαν να είναι ένα μέσο διατήρησης μιας θέσης εργασίας που αντανακλά κραβώς μια ιδιόμορφη κατάσταση ισορροπίας μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ε, ζωής ε, κάποιε ιδιαιτερότητε εδώ. Αλλά θα πρέπει βέβαια να καταχειρώνονται και τα κοινωνικά δικαιώματα των ε, μισθωτών που θα πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο με εκείνους τους εργαζόμενους που δουλεύουν με κανονικές συμβάσεις. Βεβαίω, λέγοντα όλα αυτά, θα πρέπει να σκεφτούμε τι νέε μορφέ κοινωνικού διαλόγου και είναι ουσιώδε εδώ να έχουμε τον διάλογο αυτό με τα συνδικάτα, τα οποία γνωρίζουν καλά την εργασία των μισθωτών και που θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε όλες τις διαδικασίες χάραξης κοινωνικής πολιτικής. Ιδού λοιπόν αυτά που θέλω να σας πω εισαγωγικά. Δεν ξέρω αν θέλετε να πω κάποια πράγματα για τις τροπολογίες που κατέθηκαν από τους συναδέλφους ή να προηγηθεί η συζήτηση και να απαντήσω μετά. Δεν ξέρω. Νομίζω θα ήταν χρήσιμο να ξεκινήσουμε συζήτηση και να Περιμένουμε να δούμε τι σχόλια θα προκύψουν και κατόπιν μπορούμε να επανέλθουμε στις ε, τροπολογίες. Πρώτος και καλύτερος ο κύριος Κοφεράτη. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την ε, συνάδελφο που συνέταξε την πρόταση αυτή. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση και όχι μόνο ενδιαφέρουσα από την άποψη της ανάλυσης της ε, ισχύουσας κατάστασης, αλλά περιλαμβάνει και κάποιες ε, δηλώσεις αρχής που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικές και να μπορούμε να εργαστούμε, συνεργαστούμε θετικά συμπληρώνοντας το κείμενο. Γι' αυτό το λόγο θα περιοριστώ στο να επιμείνω σε κάποιες πτυχές που υπάρχουν στο κείμενο και που θεωρώ είναι σημαντικές. Όταν γίνεται λόγος για άτυπες συμβάσεις, είναι απαραίτητο να θεωρήσουμε δεδομένο ότι το σταθερό σημείο αναφοράς είναι το, η σύμβαση ορίστου χρόνου που συνοδεύεται από διάφορες άλλες μορφές. Αυτές οι διαφορετικές μορφές θα πρέπει να αποκρίνονται σε ορισμένου συγκεκριμένους κανόνες και όχι να χρησιμοποιούνται μόνο για να περιορίζεται το κόστος μιας εταιρείας. Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό να έχουν οι άνθρωποι τη δυνατότητα να επιλέγουν και την δική τους ιδέα για τη ζωή ανάμεσα από διάφορες ε, λύσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που προτιμούν να εργάζονται με ένα συγκεκριμένο, για ένα συγκεκριμένο σύμβαση ορισμένου χρόνου με διαφορετικούς όρους δηλαδή από ότι οι πατεράδες τους ή οι παππούδες τους. Έπειτα, το, η σύμβαση ε, του χρόνου όπως και η άτυπη εργασία θα πρέπει να θεωρούνται ως ευκαιρίες που ε, περιέχουν και ποιότητες, ποιοτικά στοιχεία. Η αξιοπρεπής εργασία και εργασία η ποιοτική ισχύει για όποια μορφή εργασίας και να μιλάμε. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό το μέσο της κατάρτισης που επιτρέπει όχι μόνο το πέρασμα από τη μια μορφή στην άλλη, αλλά επιτρέπει το εσωτερικό κάθε μορφής να ενημερώνεται κανείς επαγγελματικά. Γιατί με τα όσα μάθανε κανεί στο σχολείο όταν ήμουν εγώ μικρό, μπορούσε να δουλεύει για 20 χρόνια ήσυχο. Ενώ τώρα οι σχολικές ε, γνώσεις εξαντλούνται σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ένα άλλο σημείο επίσης. Οι ευρωπαϊκές οικονομίες ε, κάποιες φορές επιβαρύνονται και καθορίζονται από την παράνομη εργασία. Οι μορφές παράνομης εργασίας επίσης διαφέρουν μεταξύ τους. Μιλάμε για την ε, συγκαλυμμένη τη μαύρη, συγκαλυμμένη μάλλον εργασία που βασικά αφορά τους ξένους και πάει μέχρι την μαύρη αγορά, μαύρη αγορά που σημαίνει ότι εργάζεται κανείς χωρίς σύμβαση εργασίας και θα πρέπει να μπορέσουμε να αποθαρρύνουμε αυτές τις μορφές εργασίας τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τον ανταγωνισμό γιατί εκεί όπου υπάρχει παράνομη εργασία αλλάζουν οι σχέσεις ανάμεσα στις εταιρείε. Γι' αυτό δεν νομίζω πως αρκεί να έχουμε στη διάθεσή μας μια πολλαπλότητα μέσων, αλλά πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες πολιτικές που έχουν στόχο ε, την ε, διαφορά, την αντιπαράθεση ανάμεσα στα νόμα και στα απαράνομα, στις παράνομες μορφές εργασίας. Και έπειτα, η ίδια λογική ισχύει και για τα δικαιώματα. Τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων θα πρέπει να είναι καθολικά και να αναγνωρίζονται ως καθολικά. Τόσο για όποιον έχει σύμβαση ορισμένου χρόνου, όσο και όποιο, για όποιον επιλέγει οποιαδήποτε μορφή άτυπης εργασίας. Έτσι ώστε να μην υπάρχει το δίθεν ατυπικό που αποκαλείται έτσι, αλλά είναι απλώς ένα παραθυράκι για να μειωθεί το κόστος εις βάρος των ατόμων. Το βασικό επιχείρημα που αναφέρεται σε όλες τις χώρες τώρα είναι αυτό. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και την αξία της συλλογικής σύμβασης. Μίλησε για ατομικά δικαιώματα, αλλά είναι προφανές πως η συλλογική σύμβαση είναι ένα συλλογικό μέσο που είναι εξίσου σημαντικό. Η δυνατότητα να παρουσιαστεί κανείς ελεύθερα δεν είναι μόνο ένα στοιχείο ε, πολιτισμού και της ε, ιδιότητας του πολίτη, όχι, είναι και ένα στοιχείο το οποίο λειτουργεί κατά του ντάμπινγκ. Τώρα, τις τροπολογίες που έχω υποβάλει και τις άλλες που υπέβαλαν διάφοροι συνάδελφοι, καθορίστηκαν από την πρόταση των, προτάσεών σας. Δηλαδή παρουσιάσατε τις ε, θέσεις σας με ανοιχτά παράθυρα, ε, επιτρέποντας και στους υπόλοιπους να συμβάλλουν για ένα τόσο λεπτό θέμα όπως αυτό. Η κυρία Στένμπρουκ. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Όπως ε, ήδη είπα στο προηγούμενο θέμα της ημερησίας διάταξης, με ενδιαφέρει ε, να διατηρήσουμε τον στόχο όσον αφορά τις ε, συνθήκες εργασίας. Να μην ξεφύγουμε από τον και εδώ θα πρέπει να λάβουμε κατάλληλα μέτρα και γι' αυτό έχουμε υποβάλει τροπολογίες οι οποίες αναφέρονται στις εργασιακές ε, σχέσεις και στόχο έχουν να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα και να καταπολεμηθούν οι ανισορροπίες ανάμεσα σε άτυπες και τυπικές συμβάσεις. Πάντα πρέπει να καταδικάζουμε τις δυσανάλογες ε, συνθήκες εργασίες που προκύπτουν από άτυπες συμβάσεις. Ε, μας ε, ενδιαφέρουν όχι μόνο οι ε, ευκαιρίες φροντίδας των παιδιών αλλά και οι ώρες εργασίας που να επιτρέπουν μια κανονική οικογενειακή ζωή και επίσης κάποια μέτρα επιτρέπεται να καταργούνται μόνο όταν δεν εξυπηρετούν την προστασία του εργαζομένου. Ευχαριστώ πολύ κύριος Κρίστενσεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι αν θέλουμε η ισορροπημένη flexicurity χρειάζεται ε, μεγάλη ευελιξία στην αγορά εργασίας αλλά και κοινωνική ε, ασφάλεια. Και θα πρέπει να υπάρχει υποστήριξη σε περίπτωση που μείνει κάποιο άνεργο ε, και να μπορεί να ζήσει από αυτήν, να μην πρέπει να καταλήψει το σπίτι του. Θα πρέπει να λαμβάνει κανεί μετεκπαίδευση ώστε να μπορεί να κινηθεί στην αγορά εργασία, να μεταφερθεί σε άλλου τομεί σε περίπτωση που πάψει να υπάρχει ο τομέα στον οποίο εργαζόταν κανεί και ε, πρέπει να υπάρχει επίσης ενεργός ε, πολιτική εργασίας, να υπάρχουν ε, μεμονωμένα σχέδια δράσης για κάθε άνεργο, ώστε αυτός να μεταφέρεται σε κατάλληλο μέρος. Εάν υπάρχουν αυτά όσον αφορά την ασφάλεια, τότε θα έχουμε ευελιξία στην αγορά εργασίας. Έτσι λειτουργούν τα πράγματα στη Δανία, επειδή έχουμε επενδύσει τόσα χρήματα στην πολιτική της αγοράς εργασίας. 6,5% περίπου του ΑΕΠ δαπανούμε για την πολιτική της αγοράς εργασίας και γι' αυτό έχουμε πολύ ευέλικτο εργατικό δυναμικό. Στην Ευρώπη όμως αυτό που είδαμε στις αγορές εργασίας είναι ότι προσλαμβάνεται κανείς με βάση ένα σωρό περίεργες συμβάσεις όπου εργάζεται κανείς υπό κακές συνθήκες και με κακή αμοιβή. Είναι σημαντικό αυτές οι μορφές διορισμού να μην χάνονται σε κάποιες γκρίζες ζώνες. Ε, έχουμε ένα σωρό οδηγίες, συμβάσεις για για μερικό, μερική απασχόληση ε, για πρακτική άσκηση κλπ. Ε, θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να μην ε, προσλαμβάνεται κανείς με βάση περίεργες συμβάσεις υπό κακές συνθήκες, εργατικές συνθήκες και θα ήθελα αυτό να το κοιτάξει η συγγήτρια. Επίση, σημαντικό είναι την ευελιξία με ασφάλεια, το flexicurity, να μην το χρησιμοποιήσουμε για να λύσουμε τα πάντα. Διότι ε, παρουσιάζεται ω γενική λύση για το μέλλον. Θα πρέπει όμω να ξεκινήσω λέγοντα ότι αν δεν έχει κανεί την, την απαραίτητη κοινωνικού ασφάλεια, το μοντέλο flexicurity, η ευελιξία με ασφάλεια, δεν θα λειτουργήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ο κύριος Πακ. Vorsitzende. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την αναγνώρισή μου της έκθεσης γιατί η έκθεση δεν ε, θίγει μόνο πολλά θέματα αλλά δίνει και πολλά ερεθίσματα σε σχέση με τη βελτίωση των θέσεων απασχόλησης. Γενικά έχω όπως και προλύσασα την άποψη ότι θα πρέπει να είναι ο κανόνας να έχουμε μακροπρόθεσμες συμβάσεις εργασίες. Αυτός θα πρέπει να είναι ο κανόνας, όχι κάτι που συμβαίνει τώρα στην κρίση, δηλαδή όλο και περισσότερο να έχουμε άτυπες συμβάσεις εργασίες. Τα προβλήματα είναι γνωστά ε, οι επιπτώσεις ε, στις συντάξεις, η επιδίνωση της ε, περίθαλψης κλπ, η μείωση του επίπεδου κατάρτισης, οι επισφαλείς συνθήκες υγείας και ασφάλειας στη θέση εργασίας. Εάν δούμε τι σκέφτεται η Επιτροπή σε σχέση με τις συντάξεις, πηγαίνουν ε, στο δρόμο της παρουσίασης των άτυπων συμβάσεων σαν τον κανόνα. Δηλαδή μέτρα κατάρτισης και λοιπά όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται τελικά στη συζήτηση για το συνταξιοδοτικό. Και αυτό με προβληματίζει ιδιαίτερα από τη δική μου πλευρά. Θεωρώ ότι και η καταπολέμηση της παράνομης εργασίας είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει πολύ περισσότερο και αυτό, γιατί αυτό δεν έχει μόνο ανθρώπινες επιπτώσεις, επιπτώσεις εργαζόμενους, αλλά έχει και επιπτώσεις στα συστήματα ασφάλισης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θεωρώ ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτεί κανείς την κρίση για να ενισχύσει την μετάβαση από κανονικές άτυπες συμβάσεις εργασίας για να υπονομεύσει το κοινωνικό δίκαιο στην Ευρώπη. Νομίζω ότι διάφορα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί στην παρούσα συγκυρία λόγω της κρίσης ούτε ώστε να για να μην ε, διολυστήσουν ακριβώς οι εργαζόμενοι σε αυτές τις άτυπες ε, συμβάσεις και τις επισβαλείς συνθήκες εργασίας. Θα πρέπει να εμποδίσουμε αυτό το φαινόμενο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα του τι θα το ποιο θα πρέπει να είναι ο στόχο αυτή τη έκθεση κατ' ουσία. Έχω την άποψη ότι ο στόχο αυτή τη έκθεση θα πρέπει να είναι μια δήλωση αυτή τη Επιτροπή. Να πούμε δηλαδή ότι οι συμβάσει του χρόνου είναι οι κανονικέ συμβάσει εργασία. Ε, νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο είχε παρουσιαστεί πολύ ξεκάθαρα στην αρχή μια συνεδρίασή μα, όταν είπαμε ποια είναι η κατάσταση η οποία δημιουργείται όταν οι ε, προσωρινές ε, συμβάσεις εργασία τελικά γίνονται ο κανόνας και με τον τρόπο αυτό υπονομεύονται τα κοινωνικά συστήματα και πλέον οι συντάξει δεν μπορούν να παρέχουν απολύτω καμία ασφάλεια. Και θα ήθελα να προσθέσω εδώ ένα άλλο στοιχείο το οποίο θα συζητήσουμε περισσότερο από ευκαιρία τη δική μου έκθεση. Το γεγονό ότι εάν υπάρχουν μόνο περιορισμένε ε, συμβάσει εργασία, περιορισμένο χρόνο δηλαδή, τότε θα βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου μια κοινή ευθύνη μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη θα πρέπει ότι η κοινή αυτή πρέπει να επιληφθεί από κοινού και θα πρέπει να υπάρξουν ε, ευκαιρίες κατάρτισης στη θέση εργασίας. Νομίζω ότι έχουμε τα τεχνικά μέσα να δημιουργήσουμε νέες θέσεις ε, απασχόλησης, αλλά δεν έχουμε τους ειδικευμένους εργαζόμενους οι οποίοι δεν είναι διατεθειμένοι να μπουν σε συμβάσεις περιορισμένου χρόνου αλλά θέλουν μόνιμες συνθήκες εργασίας. Νομίζω ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουμε στοιχεία που αφορούν τα ζητήματα της συνοχής στην πολιτική της απασχόλησης γιατί υπάρχουν περιοχές πολύ φτωχές όπου ε, οι επισφαλείς συνθήκες εργασίας γίνονται ο κανόνας. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει πολύ περισσότερο και έχω την άποψη η βασική τάση η οποία αναφέρεται σε αυτή την έκθεση εύκολα παρερμηνεύεται δηλαδή ε, εμφανίζονται οι άτυπες συμβάσεις σαν να είναι η μόνιμη λύση ε, για το μέλλον. Νομίζω ότι θα πρέπει να απορρίψουμε ξεκάθαρα αυτή την τάση, επαναλαμβάνοντας ότι ο κανόνας θα πρέπει να κατησχύσει ότι οι τυπικές συμβάσεις εργασίας, οι συμβάσεις αορίστου χρόνου, είναι η φυσιολογική συνθήκη εργασίας. Ευχαριστούμε, κύριος Όρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την ε, Πασκάλ Γκρουνή για την εξαιρετική της εργασία. Είναι πολύ σημαντική η έκθεση αυτή. Τίνω να διαφωνήσω με κάποιες από τις παρατηρήσεις που άκουσα από τους συναδέλφους. Δεν έχω δει όλου την αίσθηση ότι πρόκειται μόνο για ε, ευχολόγια. Το, το, ίδιο το κείμενο φων, μιλάει για τις ε, συμβάσεις αορίστου χρόνου, όμως ε, ο κόσμος αλλάζει. Βρισκόμαστε σε, σε πλαίσιο παγκόσμιου ανταγωνισμού είτε μας αρέσουν ε, τα, οι συμβάσεις ε, με σταθερούς όρους ή όχι, υπάρχουν όλο ένα και περισσότερο άτυπες μορφές εργασίας και αυτές οι, ε, τα άτυπα, οι άτυπες συμβάσεις εργασίας εξαπλώνονται όσο, όσο πάει και περισσότερο. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι η έκθεση αυτή περιγράφει την κατάσταση χωρίς να την κρίνει. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βάλουμε μια κάποια τάξη σε αυτόν τον κόσμο γιατί αυτή τη στιγμή οι ευθύνες ε, δεν ορίζονται, ε, το βάρος ε, δεν μοιράζεται, κανείς δεν ξέρει ποιος είναι υπεύθυνο γιατί όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας βρισκόμαστε σε ένα no man's land, σε μια τελείως εφαία ζώνη όπου ε, ισχύει η δύναμη, το δίκαιο του ισχυροτέρου. Εγώ δεν θέλω να κρίνω την άτυπη εργασία, αν είναι καλή ή κακή, αν είναι αυτό που θέλουμε ή αυτό που απευχόμαστε, αλλά καλύτερα είναι να δούμε ε, κάτι, να δούμε τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτές τις μορφές, ποια είναι τα δικαιώματα τους και ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους, όπως κάνουμε και για τις υπόλοιπες συμβάσεις εργασίας, τις πιο συνηθισμένες, τις πιο φυσιολογικές. Οι κανόνες για την απασχόληση περιγράφουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ανθρώπων που απασχολούνται σε κάποιες ε, μορφές, με κάποιες συγγνώμη, μορφές συμβάσεων και το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε με τις άτυπες μορφές, είτε μας αρέσει είτε όχι να πρέπει να συνηθίσουμε αυτού του είδους ε, τις άτυπες μορφές εργασίας, γιατί πολλές από τις θέσεις απασχόλησης που χάθηκαν τους περισμένους μήνες, ποτέ δεν πρόκειται να επανέλθουν. Και πολλοί κόσμος που ξαναβρίσκει δουλειά, θα βρει δουλειά με άτυπη μορφή. Πολύ σημαντική έκθεση λοιπόν, γιατί είναι πραγματικά μια έκθεση με μακρόπνοη και προσπαθεί να προβλέψει πώς θα καλύψουμε τέτοιο είδους μορφές εργασίας. Ο κύριος Μάν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι ο κύριος Ερία αναφέρθηκε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Κυρία Γκρίνη, σας ευχαριστούμε πολύ για την καλή έκθεση. η οποία δεν θέλει να λάβει απόφαση που να ισχύει για όλους. Έχουμε διάφορες βάσεις, διαφορετικά περιθώρια δράσης. Ε, πιστεύω πάντως ότι είναι πολύ καλή βάση και το γεγονός ότι ε, έχουν υποβληθεί 200 ε, τροπολογίες δεν σημαίνει ότι είναι αδύναμη η έκθεση. Δείχνει την πρόθεση να εργαστούμε περισσότερο πάνω στο θέμα και γι' αυτό είμαι ευγνώμων. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα της πλήρους απασχόλησης. Ναι, θα ήταν πολύ ωραίο αυτό, αλλά τι θα γίνει αν σε πολλούς τομείς δεν είναι δυνατή η πλήρης απασχόληση, διότι οι κατάσταση αγορές είναι ανασφαλής, δεν ξέρουμε ποιες επιχειρήσεις μπορούν να επιβιώσουν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ξέρουμε ποια, ποιοι παράγοντες υπάρχουν που να μπορούν να διασφαλίσουν την απασχόληση επειδή ο κοινωνικός διάλογος δεν είναι σε όλα τα κράτη-μέλη τόσο επιτυχής όσο θέλουμε. Ε, τι θα γίνει τότε. Ε, να μην ε, έχουμε την πλήρη απασχόληση ως σύνθημα, να σκεφτούμε ε, πού υπάρχουν διαφορετικές ε, συνθήκες εργασίας, που υπάρχουν ευέλικτες συνθήκες εργασίας, ώστε οι άνθρωποι να έχουν συμβάσεις τις οποίες να μπορούν να δεχτούν. Να νιώθουν ότι είναι μέρος ε, μιας ανάπτυξης ε, η οποία ε, είναι βιώσιμη στο μέλλον. Πολύ σωστά η κυρία Σρέτερ αναφέρθηκε σε μια περιφέρεια όπου ο κόσμο είναι ευγνώμων που αν μπορεί να βρει δουλειά και ότι οι εργοδότε αυτό το εκμεταλλεύονται. Δεν μπορούμε να έχουμε κάτι τέτοιο. Φυσικά είμαστε υπεύθυνοι για τι συνθήκε πλαίσιο που θα δημιουργήσουμε ώστε η σύμβαση αορίστου χρόνου να είναι ε, η συνήθι σύμβαση. Ο κόσμος θα πρέπει να μπορεί να διαλέξει. Χρειαζόμαστε όμως μία έκθεση ε, που να μην ε, αναφέρει απλά στόχους, να αναφέρει και την πραγματικότητα που ισχύει. Ευχαριστώ τον Όλε Κρίστενσεν. Είχαμε μια εξαιρετική έκθεση από αυτόν. Μάθαμε από αυτόν τι σημαίνει η ευελιξία με ασφάλεια. Όλα αυτά ισχύουν. Πέρα από την ευελιξία θέλουμε και ασφάλεια. Και ακριβώς γι' αυτό εργαζόμαστε υπό μεγάλη πίεση. Θα πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε, όχι να κοιτάξουμε μόνο τις επιθυμίες μας και γι' αυτό ε, θα πρέπει οι κοινωνικοί εταίροι να μπορούν να εργαστούν, να είναι ισχυροί, θα πρέπει να μπορούν να πετύχουν ε, ε, ε, ε να συνάψουν κοινωνική σύμβαση και δεν θέλουμε κοινωνικούς εταίρους που να είναι αντίπαλοι. Δεν θέλουμε δηλαδή να, να έχουμε μόνο ένα τομέα, το κράτος που είναι πάρα πολύ ισχυρό και οι άλλοι να είναι αδύναμοι. Και επίσης ε, στην τελευταία ε, ε, θητεία είχαμε μια πολύ καλή εμπειρία. Θα πρέπει να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στην νόμιμη και στην παρανόμη απασχόληση. Και είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση στην Ολομέλεια κατά του τότε Επιτρόπου Σπίτλα που ήταν απομονωμένος στις θέσεις του. Σε κάποια κράτη-μέλη έχουμε την αστυνομία και το τελωνίο που θέλουν απλά να ανακαλύψουν τους τους ε, παράνομους εργαζομένους και ε, αυτός είπε ότι ε, αυτό είναι παραβίαση της ελεύθερης κινητικότητας. Όχι, χρειαζόμαστε δικαιοσύνη, χρειαζόμαστε λογικούς ελέγχους. Εάν μπορέσουμε να τα κάνουμε αυτά καλά, τότε πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε και έτσι θα δώσουμε μια ευκαιρία στην οικονομία της αγοράς. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε συμφωνήσουμε πάνω σε πολλές από τις τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χέντελ. Ο συνάδελφος Μαν στη συζήτηση για τις κατευθύνσεις γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης με παρεξήγησε Κάτι θα σκεφτώ και εγώ για το δικό σου όνομα. Θα ήθελα όμως να πω ότι έχει δίκιο όσον αφορά ένα σημείο. Είναι πολύ καλή βάση η έκθεση της κυρίας Κρούνη, αλλά ακριβώς ε, αυτό είναι το θέμα, αγαπητέ συνάδελφε Μαν. Εάν η Κομισιόν τουλάχιστον θα μπορούσε να αναγνωρίσει ε, ποια είναι η βάση πολλών αποφάσεων εδώ του Κοινοβουλίου, Εάν το έκανε αυτό η Κομισιόν, τότε δεν θα είχαμε ε, τέτοιε κατευθυντήρε γραμμέ για την απασχόληση, θα ήταν πιο συγκεκριμένε. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει. Στην έκθεση τη κυρία Γκρούνη έχουμε μια καλή βάση. Θα πρέπει όμω να συμφωνήσουμε πάνω σε άλλα θέματα. Πιστεύω ότι μπορεί να βελτιωθεί η έκθεση αυτή και μάλιστα αρκετά. Και συνάδελφε Μαν, το θέμα εδώ δεν είναι να έχουμε την πλήρη απασχόληση ως σύνθημα θέλουμε σε, άλλους, σε άλλα μέρη του κόσμου οι άτυπες ε, συμβάσεις είναι ο κανόνας και η σύμβαση ε, απεριόριστου χρόνου ε, έχει καταργηθεί. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Θέλουμε η σύμβαση αορίστου χρόνου να είναι ο κανόνας. Δεν έχω αντίρρηση ο κόσμος να έχει άτυπες συμβάσεις αν το θέλει. Ε, επί 25 χρόνια βλέπω κάτι τέτοιο στον τομέα των υφασμάτων, για παράδειγμα, όπου προσπαθούμε να ε, εισάγουμε την ευελιξία. Αλλά γενικά στον οικονομικό τομέα διαπιστώνουμε ότι υπάρχει περισσότερη ανασφάλεια από ό,τι είναι απαραίτητο και περισσότερη και ότι απαιτείται περισσότερη ευελιξία από τους εργαζομένους ε, από ό,τι τους προσφέρεται η ασφάλεια. Και αυτό θέλουμε να αντιμετωπίσουμε στα πλαίσια της έκθεσης αυτής. Ο συνάδελφος ε, Ρή αναφέρεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων. Ε, αλλά συνάδελφε Ρή, ε, υποχρεώσεις ναι, αλλά δικαιώματα δεν έχουν Διότι μπορεί στο χαρτί να λέει ότι ένα εργαζόμενο μπορεί να. ένα ελεύθερο επαγγελματία, για παράδειγμα, ή ε, κάποιο που, είναι, ε, ε, που έχει προσληφθεί για περιορισμένο χρόνο. Εάν απαιτήσει τα δικαιώματα που υπάρχουν στη σύμβασή του, δεν θα τον ξαναπροσλάβουν. Και δεν αναφέρομαι στο εισόδημα, αναφέρομαι στο καθεστώς των εργαζομένων αυτών. Και πιστεύω ότι αυτό Μπορούμε να το βελτιώσουμε στην έκθεση αυτή της κυρία Γκρούνη. Υπάρχει μια σειρά τροπολογιών, ωστόσο, συνάδελφε Μαν, δεν θα ήθελα να επανέλθω σε αυτά που ε, διατύπωσαν ε, το, ήδη το 2007 οι ε, Υπουργοί Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρώπης. Λένε ότι τα καλά δικαιώματα είναι η κοινωνική προστασία, η προστασία υγείας για τους εργαζομένους, δίκαιες συνθήκες εργασίας και διάφορα άλλα πράγματα, διαβάζει πολύ γρήγορα ο μιλητής, που είναι απαραίτητα για τις καλές συνθήκες των εργαζομένων και των πολιτών. Ναι, είναι σημαντικό το ότι ε, ήδη τότε είχαν φτάσει εκεί οι Υπουργοί, αλλά θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην οπισθοχωρήσουμε και για να μην οπισθοχωρήσει και η Κομισιόν. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ναι, έχω κι εγώ κάποιες παρατηρήσεις. Από τη συζήτηση φαίνεται να προκύπτει ότι εάν η άτυπη σύμβαση ε, είναι επιλογή, τότε δεν έχει κανένα αντίρρηση. Έχει αντίρρηση όταν ε, επιβάλλεται αυτή και γι' αυτό έχω υποβάλει κάποιες από τι τροπολογίε μου για τους ανεξάρτητους ε, απασχολούμενους, διότι πολύ συχνά αυτοί ξεχνιόνται στην εξίσωση. 5 με 10% των απασχολούμενων εργάζονται ως ανεξάρτητοι και το επιλέγουν αυτό όχι ως μικρές, επιχειρήσεις, ως μικρές επιχειρήσεις, αλλά ως αυτοαπασχολούμενοι. Και δεν φαίνεται να ε, ε, καλύπτονται από την νομοθετική διαδικασία και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και ε, από εκεί προκύπτουν πολλές από τι τροπολογίε μου. Άλλο θέμα είναι ότι κάποιοι επιλέγουν άτυπε συμβάσει ή προσωρινή εργασία επειδή έχουν να φροντίσουν ε, παιδιά ή άλλους ανθρώπους. Ε, και ε, σημαντικό είναι να μην καταργήσουμε την, τις άτυπες συμβάσεις για τους ανθρώπους που τις χρειάζονται. Μπορεί κάποιος να φροντίζει τα παιδιά του και να είναι επιλογή αυτό. Δεν είναι όλες οι άτυπες συμβάσεις καταχρηστικές και αυτό είναι σημαντικό. Φυσικά κάποιες είναι, αλλά θα και θα πρέπει να φροντίσουμε να τις περιορίσουμε όπως και την αδήλωτη εργασία αλλά δεν θα πρέπει να φύγουμε από εδώ με την ιδέα ότι ό,τι είναι άτυπο είναι κακό ενώ οι τυπικές συμβάσεις είναι καλές διότι υπάρχουν ε, άνθρωποι οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευση ε, και ε, στι τυπικέ συμβάσει. Εάν λοιπόν είναι επιλογή η άτυπη σύμβαση, τότε εντάξει. Το άλλο θέμα για το οποίο ε, έχω υποβάλει τροποποίηση Τροπολογίε είναι οι συλλογικέ διαπραγματεύσεις, διότι δεν έχουν όλα τα κράτη-μέλη ε, σχετική παράδοση. Δεν θα πρέπει λοιπόν να το ε, θεωρήσουμε αυτό προϋπόθεση. Ναι, όπου υπάρχει σχετική παράδοση, οι συλλογικέ διαπραγματεύσεις ε, είναι κάτι πολύ καλό και θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει. Αλλά σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική παράδοση και να μην πιστεύουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν τις ίδιες παραδόσεις και ότι θα πρέπει όλοι να φορέσουμε σουρλομανδία ή κορσέ τέλο πάντων για να ακολουθούμε μόνο μία οδό για την σύναψη εργασιακών συμβάσεων. Ε, και, να μην υποχρεώσουμε δηλαδή τα κράτη-μέλη, οι μεγάλοι κοινωνικοί εταίροι να συμμετέχουν στην διαδικασία, διότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Αλλά κυρία Γκρουίνη, σας ξαναδίνω το λόγο για να αναφερθείτε σε τροπολογίες που έχουν υποβάλει συνάδελφοι ή για να απαντήσετε στα σχόλια που έγιναν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση και κατέθεσαν και τις τροπολογίες τους. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σχεδόν σε όλους. Κύριε Κοφεράτη, καταθέσετε επίσης πολλές τροπολογίες και κάθε φορά ε, ε, ε, θέλετε να δείξετε θα πρέπει να προσθεθεί η κρίση, να επισημανθεί η κρίση. Εγώ αναφέρω την κρίση νομίζω δύο ή τρεις ε, φορές καθώς και στην ιδεολογική έκθεση αλλά θεωρώ ότι η έκθεση αυτή θα πρέπει να επικεντρωθεί στην κρίση γιατί οι τυπικές συμβάσεις υπάρχουν και σε άλλες ε, ε, οι άτυπε συμβάσει υπάρχουν και σε άλλε περιόδου. Δεν θα πρέπει να αναχθούν αποκλειστικά στην κρίση. Θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω ότι οι συμβάσει αριστοδιάρκειας ε, ήταν ο κανόνας. Μιλήσατε για την διαβίου μάθηση, την αναφέρω επίσης και τη σημασία των συλλογικών ε, διαπραγματεύσεων, συλλογικών συμβάσεων. Υπάρχει μια τροπολογία την οποία δεν κατάλαβα πολύ καλά του κ. Ρή και υπάρχει επίσης ε, μια άλλη τροπολογία που αφορά τη μοιρασιά ανάμεσα στην οικογενειακή και την επαγγελματική ζωή. Και ίσως αυτές οι άτυπες συμβάσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια επιλογή για αυτά τα άτομα που θέλουν να μοιράσουν ε, την επαγγελματική και την προσωπική του ζωή με αυτόν τον τρόπο. Ε, κυρία Κρόνερ, είπατε ότι θα πρέπει να καταδικάσουμε τις άτυπες συμβάσεις. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να τις καταδικάζουμε. Πιστεύω ότι θα πρέπει να τις πλαισιώσουμε. Αλλά είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει και ορισμένε φορές συνιστά μια επιλογή. Αλλά αν τις πλαισιώσουμε σωστά, δεν ξέρω ήταν και ένα πρόβλημα μετάφρασης, ή αν τις πλαισιώσουμε σωστά, και νομίζω ότι αυτός είναι ένας στόχος της έκθεσής μου, ε, δεν θα δούμε να υπάρχουν εντελώς ε, ε, συμβάσεις που οδηγούν τους εργαζόμενους σε μεγάλες ε, δυσκολίες σε σχέση ακριβώς με την κοινωνική τους προστασία. Κύριε Κρίστενσεν, μιλήσατε ε, για το ζήτημα της ε, επαγγελματικής ε, ζωής που παλιά ήταν ε, κάτι που διαρκούσε μια ζωή, η ίδια δουλειά. Σήμερα θα διαρκέσει μια ζωή. Σήμερα αλλάζει κανείς πολλές φορές επάγγελμα. Συνεπώς η διαβίου κατάρτιση είναι σημαντική για ανθρώπους που εργάζονται μεν, αλλά κάποια στιγμή μπορούν να έρθουν αντιμέτωποι με κάποια αλλαγή ή εξέλιξη και θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να είναι σε θέση να διατηρήσουν μια θέση εργασίας, να στραφούν κάπου αλλού. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Και η έκθεση αυτή θα πρέπει πάντα να συμπλάνει αυτό το θέμα της ε, διαβίου εκπαίδευσης. Μιλήσατε επίσης για τις ε, επιχειρήσεις ε, για μια ψευδοανεξαρτησία δεν είναι δυνατόν να είναι κανείς ε, είτε ανεξάρτητος επαγγελματίας είτε μισθωτός ή το ένα και το άλλο ταυτόχρονα. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Κύριε Μπάρτ, μιλήσατε για το θέμα της κοινωνικής προστασίας και είμαι πολύ του σύμφωνη μαζί σας. Πέρσι στη Γαλλία, σε σχέση με τους ανθρώπους που φεύγουν από τις επιχειρήσεις, ε, ε, θεσπίστηκε ένα σύστημα βάσει του οποίου μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να εποφελούνται από ένα επικουρικό ε, ταμείο ε, περίθαλψης για αρκετούς μήνες αυτή τη στιγμή ε, χάνουν τη θέση τους εργασίας. Νομίζω ότι αυτή είναι η σκέψη την οποία πρέπει να στηρίξουμε και τις άτυπες συμβάσεις. Και αληθεύει βέβαια όσα είπατε για τις συντάξεις. Στην έκθεσή μου όταν μιλάω για κοινωνική προστασία ενώ όλα αυτά τα θέματα και βεβαίως και τις αποζημιώσεις των ανθρώπων αυτών όταν βρίσκονται σε ανεργία και τα επιδόματα. Ε, Βεβαίω δεν θα πρέπει κανεί να εκμεταλλευτεί την κρίση για να πολλαπλασιάσει ανεξέλεγκτα τι άτυπε συμβάσει. Αυτό είναι το Η ίδια η κρίση ε, βεβαίω έχει προσθέσει ε, κάποιες ε, δυσκολίες στις άτυπες συμβάσεις που ήδη προϋπήρχαν. Εγώ ήμουν σε μια επιχείρηση μεταφορών πριν από τρία ή τέσσερα χρόνια οι οδηγοί που ήταν πλήρως απασχολούμενοι ήθελαν να έχουν προσωρινή εργασία, ήταν δική τους επιλογή γιατί ήταν καλύτερα αμοιβόμενοι. Σήμερα κάτι τέτοιο δεν ισχύει πλέον γιατί ακριβώς υπάρχει ένα πρόβλημα έβρεσης, εξέβρεσης θέσης εργασίας. Ε, κυρία Σρέτερ, Μιλήσατε για τις συμβάσεις αορίστου διάρκειας ε, που ήταν ε, ο κανόνας στο παρελθόν και που θα πρέπει να παραμείνει ο κανόνας. Όταν έχουμε επισφαλείς συμβάσεις ακόμα στο επίπεδο των επιχειρήσεων, δεν νομίζω ότι μπορούν να αποτελέσουν μια λύση, γιατί τα κίνητρα εδώ δεν είναι τα ίδια. Η συνεχής κατάρτιση, βεβαίως συμφωνώ μαζί σας, οι συντάξει βεβαίως έχετε δίκιο και ο στόχος εδώ το επενθυμίζω είναι να πλαισιώσουμε κατάλληλα αυτές τις συμβάσεις που ούτως ή άλλως υπάρχουν. Ανρί, σε ευχαριστώ για την ε, υποστήριξή σου, για τη βοήθεια που μου έδωσες για αυτή την έκθεση και λες ότι θα πρέπει να σκεφτούμε για τις μελλοντικές προσλήψεις στη μετακρίση εποχή μετά την κρίση εποχή. Ε, θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, γιατί οι επιχειρήσεις ανησυχούν λόγω αυτής ακριβώς της κρίσης ε, δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά μιας μελλοντικής αγοράς. Όταν υπάρξει μια ανάκαμψη στην αρχή θα ισχύσουν αυτές οι άτυπες ε, συμβάσεις. Όπως σας είπα, πρέπει να τις πλαισιώσουμε πιο κατάλληλα. Ή μάλλον όχι όταν υπάρχει ανάγκαψη, όταν οι άνθρωποι αυτοί ξαναμπούν στην αγορά εργασίας υπό τις παρούσες συνθήκες. Ε, Μαν, ε, σε ευχαριστώ πολύ που μου υπενθύμησε κάποια πράγματα σε σχέση με τον ορισμό της ε, άτυπης εργασίας. Νομίζω ότι το επισήμενα ήδη, αλλά εν πάση περιπτώσει θα γίνουν κάποιοι συμβιβασμοί ε, και θα τους ε, προτείνω. Κύριε Χέντελ, ευχαριστώ. Οι τροπολογίες ήταν αρκετά απεσιόδοξες θεώρησα, αλλά στα όσα, τα όσα είπατε με βρίσκουν σύμφωνοι σε πολλά σημεία και νομίζω ότι θα μπορούμε να βρούμε ένα συμβιβασμό γιατί ο δικός μου στόχος είναι πράγματι να υπάρξει μια πλήρης απασχόληση και όλοι οι εργαζόμενοι να έχουν συμβάσει αύριστο διάρκειας. Ε, δεν είναι πολιτικός μόνον ο λόγος μου. Εγώ εργάζομαι σε μια επιχείρηση ακόμα ως διευθύντρια των ανθρώπινων πόρων. Με ενδιαφέρει άμεσα το θέμα αυτό. Όσον αφορά το κοινωνικό διάλογο, αναφέρατε του προσωρινά εργαζόμενους που δεν υποφελούνται <clears throat> από αυτή τη δυνατότητα. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο κοινωνικό διάλογο. Στη Γαλλία κατοχυρώθηκε αυτό από μια, ένα νόμο του 2008 όπου μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να συμμετάσχουν στις ε, εκλογές για την εκπροσώπησή τους. <clears throat> Και θεωρώ ότι ο κοινωνικός ε, διάλογος δεν θα πρέπει να περιστεί μόνο στη σχέση εργοδότη και μισθωτού, αλλά θα πρέπει να διευρυνθεί και στους εργαζόμενους που έχουν άλλη μορφή εργασιακής σχέσης. Κυρία Λίν, ε, δεν βρίσκω σύμφωνη οι τροπολογίες σας, γιατί όπως σας είπα, είτε κανείς είναι ελεύθερος επαγγελματίας, ανεξάρτητος, ή είναι μισθωτός. Το θέμα της flexicurity, ευελιξία με ασφάλεια, αφορά τους ε, μισθωτούς. Και σκέφτομαι ότι κάποια στιγμή στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να υπάρξει ένα κείμενο για τους ανεξάρτητους επαγγελματίες, τους ελεύθερους επαγγελματίες που θα μας επιτρέψει να προσγγίσουμε το θέμα αυτό των ψευδοανεξάρτητων επαγγελματιών. Αλλά εδώ στο δικό μου κείμενο δεν νομίζω ότι έχει τη θέση του αυτή η προβληματική. Αλλά βεβαίως θα μπορούσαμε να ξαναμιλήσουμε εφόσον το επιθυμείτε σχετικά. Υπενθυμίστε τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου και ταυτόχρονα αναφερθήκατε στις παραδόσεις της κάθε χώρας μέλους όσον αφορά το κοινωνικό διάλογο αλλά εγώ πιστεύω ότι ο διάλογος οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε επίπεδο είναι ουσιώδους σημασίας. Συνεπώς η αύξηση συμμετοχής των ε, μισθωτών ε, στις επιχειρήσεις ε, είναι σημαντική. Ευχαριστώ πολύ όλους σας και <clears throat> θα επανέλθουμε για τους συμβασμούς. Σας ευχαριστώ. Σίγουρα θα έχουμε συζητήσεις για τις τροπολογίες. 2 Ιουνίου θα γίνει η ψηφοφορία στην Επιτροπή Απασχόλησης και έπειτα θα περάσει από την Ολομέλεια του Ιουνίου. Επόμενο θέμα είναι η πρόθεση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, ενίσχυση των ε, ε, μαθητευόμενων. Και στρέφουμε στην κυρία Τερών. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για τη δουλειά τους και τις πολλές τροπολογίες. Πιστεύω ότι γενικά θα μπορέσουμε να συμβιβαστούμε πολύ πάνω στο κείμενο αυτό για τον δρόμο που θα ακολουθήσουμε. Πολλές από τις τροπολογίες ε, πιστεύω ότι ενισχύουν το κείμενο πραγματικά, ενώ άλλες ε, προτείνουν ε, μικρές ή μεγάλες τροποποίησεις στο κείμενό μου. Μπορούμε να τις συζητήσουμε κατά την συνάντηση των σκιωδών εισηγητών. Ε, να σας παρουσιάσω σύντομα το κείμενο, τα πιο σημαντικά σημεία. Ως προς το εκτιμώντας ε, όπου αναφερόμαστε στις διακρίσεις των νέων και κυρίως των νέων γυναικών. Έχω υποβάλει εγώ τροπολογία για να το ε, διευκρινίσω το σημείο αυτό. Έχουν υποβάλει και άλλοι τροπολογίες όπως η κυρία Ράφτη. Ε, βλέπω όμως να υπάρχει περιθώριο συμβιβασμού όσον αφορά το ε, σίγμα ΤΑΦ που μπορεί να είναι ε, κάπως αμφιλογόμενο, ε, κάπως επίμαχο σημείο. Αρκετοί βουλευτέ έχουν υποβάλει σχετικές τροπολογίες. Θα ήθελα να σα εξηγήσω γιατί. Συνέταξα το κείμενο με το συγκεκριμένο τρόπο. Ο λόγος που το διατυπώνω την ε, τροπολογία και αναφέρω το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Δανία δεν είναι για να δαχτυλοδεικνύουμε τις χώρες αυτές και να τις κατηγορούμε. Ήθελα να αναφέρω παραδείγματα τα οποία δεν ευνοούν τους νέους στην Ευρώπη. Σίγουρα θα μπορούσαμε να βρούμε και άλλα παραδείγματα, αλλά για να είμαι ευγενική αναφέρω και τη δική μου χώρα, διότι πιστεύω ότι είναι σημαντικό να εξετάσουμε τις με μονομένες περιπτώσεις αναφερόμαστε κυρίως στα ημερομίσθια και στα επιδόματα ανεργίας. Είναι σημαντικό ε, οι νέοι να μπορούν να έχουν μια ανεξάρτητη ζωή. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αναφερθούμε στο θέμα των ε, ελάχιστων μισθών, τη μη πρόσβαση ε, στα επιδόματα κλπ. Η κυρία Ράπτη, ο κύριο ε, Χέλμερ, η κυρία Κρίνη έχουν υποβάλει σχετικέ τροπολογίες και θα ήθελα να καταλάβω Ε, γιατί δεν θέλετε συγκεκριμένα παραδείγματα. Πιστεύω ότι μπορούμε να το λύσουμε το θέμα αυτό πάντως. Όσον αφορά την παράγραφο 1, ο κύριος Χέλμερ προτείνει διαγραφή του γεγονότος ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί μια προσέγγιση βασισμένη στα δικαιώματα. Για μένα είναι Παράγραφο κλειδί αυτή και για μένα είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούμε στα, παραδείγμα, στα δικαιώματα. Συγγνώμη. Όσον αφορά την παράγραφο 2 και τι πράσινε θέσει απασχόληση, έχω υποβάλει εγώ δική μου τροπολογία, διότι πιστεύω ότι όταν στοχεύουμε στην δημιουργία νέων θέσεων απασχόληση για του νέου θα πρέπει να ε, εξετάσουμε ποιου τομεί θέλουμε να προωθήσουμε και τι νέε θέσει απασχόληση θέλουμε να δούμε στην Ευρώπη. Νομίζω ότι μπορείτε να συμφωνήσετε με αυτό. Παράγραφο 3. Πολλέ τροπολογίε Συμφωνώ με την τροπολογία της κυρίας Ράπτη και τις προτάσεις της ε, να συμπεριλάβουμε τις επιδοτήσεις απασχόλησης ε, για τους νέους ε, καθώς και τα προγράμματα για κινητικότητα των νέων επαγγελματιών. Εγώ αναφέρω τα αποδοτικά κίνητρα που μπορεί να είναι και τα ε, ε, χαμηλά ημερομήσια. Νομίζω ότι αυτό πάντως λύνεται με τροπολογίες άλλων συναδέλφων. Παράγραφος 4, κυρία Ράπτη, ε, την συμπερίληψη του προσανατολισμού το εκτιμώ αυτό όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τη διάθεση συγκεκριμένων πόρων. βλέπω ότι αρκετά μέλη στηρίζουν αυτό και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε μια καλή λύση. Παράγραφος 6. Βρίσκω την πρόταση του κυρίου, του κυρίου Πουπάκη να επικεντρωθούμε περισσότερο στις πρακτικές πτυχές. Ε, βρίσκω την πρόταση αυτή πολύ ενδιαφέρουσα. Πιστεύω ότι αναφέρεται σε κάτι σημαντικό. Ε, η διάκριση που γίνεται είναι πολύ δύσκολη για κάποιους νέους, ιδιαίτερα αυτούς που έχουν πιο πολλές πρακτικές δεξιότητες. Θα πρέπει να συνδυάσουμε περισσότερο, ε, να συνδυάσουμε καλύτερα την πρακτική διάσταση με την διανοητική και νομίζω ότι μπορούμε να συμπεριλάβουμε την τροπολογία του κυρίου Πουπάκη στην έκθεση. Ε, παράγραφος 7. Να σας ε, εξηγήσω. Είχαμε πολλές ε, τροπολογίες εδώ έχουν να κάνουν με τα προγράμματα άσκησης. Ε, συνειδητοποιώ, καταλαβαίνω ότι δεν είναι πολύ ακριβέ το σημείο αυτό. Θα πρέπει να κάνουμε διάκριση ε, ανάμεσα στα προγράμματα άσκησης από τη μία και που είναι πρόσθετη άσκηση με την οποία βελτιώνουμε την αποσχολησιμότητα των νέων δίνοντάς τους πρακτική επαγγελματική άσκηση και γίνεται ε, ε, ε, μετά τις πανεπιστημιακές σπουδές. Δυστυχώς όμως αυτό έχει εξελιχθεί σε μια αρρύθμιστη αγορά εργασίας για νέους που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους. Μιλάμε δηλαδή απλά για φθηνό εργατικό δυναμικό. Από την άλλη έχουμε τη μαθητεία που αποτελούν ε, αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης. Για παράδειγμα στην Αυστρία, τη Γερμανία και τη Δανία έχουμε ε, το διτό σύστημα το οποίο θεωρείται επιτυχές. Το πρόβλημα στη μαθητεία είναι ότι είναι πολύ λίγες οι θέσεις μαθητείας και σε εποχές κρίσης οι επιχειρήσεις δεν προσλαμβάνουν μαθητευόμενους διότι ήδη δεν έχουν ε, πολύ κέρδος. Ε, είναι λοιπόν ένα σύστημα το οποίο είναι ευαίσθητο απέναντι στα οικονομικά σκαμπανεβάσματα. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί νέοι δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Είναι λοιπόν δύο διαφορετικά προβλήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με διαφορετικό τρόπο. Και γι' αυτό χώρισα αυτή την παράγραφο σε δύο νέε περιγράφου. Η μία έχει να κάνει με τα προγράμματα άσκηση, όπου ζητάμε ε, έναν ευρωπαϊκό χάρτη ποιότητα και ευχαριστώ τον Στίβεν Χιού για τι πολύ συγκεκριμένε ε, τροπολογίε του που, που αναφέρουν το τι μπορεί να συμπεριλαμβάνεται ε, ε, στον ε, χάρτη ποιότητας και που ζητάει από τα θεσμικά όργανα να βελτιώσουν την κατάσταση και από την άλλη το δεύτερο μέρος της παραγράφου αυτής έχει να κάνει με την μαθητεία. Θα κάνω γρήγορα επειδή ξέρω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο. Παράγραφος 8. Αναφερόμαστε στην δωρεάν εκπαίδευση στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο. Βλέπω ότι υπάρχει συμφωνία στην Επιτροπή μας και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Ε, flexicurity, ασφάλεια, παράγραφος 12. Ευελισφάλεια, όπως αναφέρεται στο κείμενο. Ε, αναφέρω εδώ πέρα τέσσερα στοιχεία, τα οποία είναι τα επίσημα στοιχεία τη Κομισιόν έχει ε, τροποποιηθεί η διατύπωση εδώ από πολλούς. Ε, θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε μήπως θέλουμε να ε, μείνουμε στο κείμενο της Κομισιόν και να τονίσουμε ότι και τα τέσσερα αυτά στοιχεία πρέπει να εφαρμοστούν και όχι μόνο το κομμάτι που αφορά την ευελιξία ή θέλουμε να έχουμε δικό μας ορισμό της ευελιξίας με ασφάλεια. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε κατά τη συνάντηση των σχετών εισηγητών ή με εισηγητών. Είμαι ανοιχτή στο θέμα αυτό. Η κυρία Χίρς συνδέει την συζήτηση αυτή με τις ε, συντάξεις και βρίσκω ότι αυτό είναι σημαντική προοπτική, είναι θετικό. Παράγραφος 15. Θα ήθελα να τονίσω ότι οι, καλύτεροι, οι καλύτερες δυνατότητες παιδικής μέρημνας ωφελούν κυρίως τις νέες ε, γυναίκες, διότι αυτές συνήθως μένουν στο σπίτι τους για να φροντίσουν τα παιδιά τους. Και γι' αυτό αναφέρομαι εδώ στις νέες μητέρες Πολλοί έχουν τροποποιήσει αυτό σε νέους γονείς, αλλά πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να ε, βρούμε μια λύση όσον αφορά την ε, η εγγύηση προς τους νέους. Ε, η ΓΚΟΕ προτείνει να, υπάρχει αυτή, να εφαρμόζεται αυτή αμέσως και όχι μετά από εξάμεινο ή τετράμινο, μάλλον θα πρέπει να το αλλάξουμε αυτό το τετράμινο, ε, αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε, μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Εγγύηση Νέων, θα πρέπει να σκεφτούμε αν είναι ρεαλιστικό να το εφαρμόσουν αυτό τα κράτη-μέλη, διότι θα πρέπει να ζητάμε κάτι χρήσιμο και εφαρμόσιμο. Δεν θέλω να προχωρήσω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Μία τελευταία παρατήρηση. Περιμένω να ακούσω από εσά τι έχετε να μου πείτε, αλλά μία τελευταία παρατήρηση. Ήμουνα στο Χέρας Τελαφοντέρα στην Ισπανία πριν δύο εβδομάδες σε μια διάσκεψη της Προεδρίας για την ανεργία των νέων. Εκπρόσωποι από όλα τα κράτη-μέλη, από οργανώσεις νέων, από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκπρόσωποι της Κομισιόν και της Ισπανικής Προεδρίας συναντήθηκαν και προσκλήθηκα επειδή νωρίτερα είχα έρθει σε επαφή με την Ισπανική Προεδρία σχετικά με τη διαδικασία αυτή και την έκθεση αυτή. Μπορώ να σας ενημερώσω ότι υπάρχει μια σαφής διαδικασία εντός του Συμβουλίου που προσανατολίζεται στην ε, ανεργία των νέων και πολύ σύντομα δύο συμπεράσματα αυτό το θέμα μεταφέρεται από την Ισπανική στη Βέλγικη και μετά στην Ούγγρικη Προεδρία. Ε, λαμβάνονται υπόψη εδώ τα συμβούλια των νέων ε, στην ε, διαδικασία λήψη αποφάσεων. Η Ισπανική Προεδρία έχει επικεντρωθεί στην κοινωνική ένταξη, η Βελγική επικεντρώνεται στην συμμετοχή και η Ουγγαρία στην δημιουργία θέσεων απασχόληση για του νέου. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και, η το δεύτερο μου συμπέρασμα είναι ότι θα πρέπει να σκεφτούμε πώ μπορούμε να συμμετάσχουμε στη διαδικασία αυτή, διότι εκείνοι εξεπλάγησαν ότι εμφανίστηκε καν κάποιο από το Κοινοβούλιο. Η σχέση αυτή λοιπόν ανάμεσα στα θεσμικά όργανα σίγουρα μπορεί να βελτιωθεί. Εγώ θα ήθελα πολύ να συνεχίσω τις επαφές, αλλά μέχρι στιγμής γνωρίζουμε πολύ λίγα για το τι γίνεται εκεί απέναντι και αυτό είναι κρίμα. Βέβαια αυτό είναι αμοιβαίο. Αυτή ήταν λοιπόν η τελευταία μου παρατήρηση. Θα ήθελα να το συζητήσω αυτό με τους κοιόδης συζητητές, ενδεχομένως και με την πρόεδρό μας κάποια στιγμή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γκρίνη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να απαντήσω σε σχέση με μια τροπολογία για διαγραφή που ενδεχομένω ε, οι συνάδελφοι βρίσκουν ε, προβληματική. Αφορά το revenu minimum d'insertion euh, στη Γαλλία. Οι Γάλλοι δεν μπορούν ε, να επωφεληθούν από, αυτό το, από αυτές τις ελάχιστες αποδοχές εάν έχουν αν είναι κάτω από 26 ετών. Υπάρχουν κάποιοι νέοι οι οποίοι δεν έχουν ε, πόρους και θα ήθελα να έχουν αυτό το επίδομα. Εγώ είμαι κατά ενός ε, τέτοιου, μιας τέτοιας βοήθειας προς τους νέους, γιατί τελικά τους κάνει να εθιστούν σε, τέτοιο, σε ένα τέτοιο είδος επιδόματος και τους εμποδίζει από την ένταξη στην αγορά εργασίας. Αυτό το οποίο θα επιθυμούσα εγώ είναι πράγματι οι νέοι να βρουν το ταχύτερο δυνατό μια θέση εργασίας ή να ξεκινήσουν μια κατάρτιση και στη συνέχεια να έχουν το δικαίωμα σε ένα επίδομα ε, εφόσον είναι άνεργοι και εκεί δεν ισχύει αυτό το όριο των 25 ετών. Ε, στη Γαλλία κάποιος ο οποίος ε, δεν κάνει τίποτα έχει τουλάχιστον αυτά τα χρήματα. Και εδώ εγώ θα ήθελα να σας πω ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο λέω ότι θα πρέπει να στρέψουμε τους νέους προς την απασχόληση, την κατάρτιση, όχι να τους δίνουμε χρήματα έτσι, γιατί θα τα πάρουν και δεν θα κάνουν τίποτα για τη ζωή τους. Ε, βεβαίως, ε, το συζητώ. Ο κύριος ε, Σέρκας ε, πρότεινε αυτό το την αλλαγή τη ροή αυτού του τμήματο. Εγώ συμφωνώ για τα υπόλοιπα. Δηλαδή μια αξιοπρεπή διαβίωση, κατάρτιση κλπ. Εγώ συμφωνώ σε όλα αυτά. Εγώ είμαι πολύ υπέρ της ε, μαθητείας ε, και εδώ υπάρχουν κάποιες επαγγελματικέ συμβάσει. Το ζητούμενο είναι να δοθεί το ταχύτερο δυνατό η δυνατότητα σε φοιτητέ ή νέου αυτής της μαθητείας. Δηλαδή να δοθεί μια θεωρητική και πρακτική ε, δυνατότητα μαθητείας. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό και θα πρέπει να ισχύσει παντού. Βεβαίω υπάρχουν, ε, το ερώτημα υπάρχουν αρκετέ επιχειρήσει που να μπορούν να ενσωματώσουν όλου του νέου. Γιατί υπάρχουν πολλοί νέοι που θα ήθελαν να κάνουν τέτοιου είδου μαθητή, αλλά δεν έχουν την ευκαιρία. Τώρα, όσον αφορά την αποζημ... της, ε, ε, τα χρήματα που παίρνει κανείς να παρακολουθεί ένα στάζ. Εδώ θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί εάν επιβάλλουμε ένα τέτοιο κανόνα αποζημίωσης, ε, υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν θα είναι διατεθειμένες να πληρώσουν για τους μαθητευόμενους, αυτούς που κάνουν τα στάζ. Βεβαίως, αν ο, αυτός που κάνει το στάζ ε, εργάζεται κανονικά, φυσικά θα πρέπει να αποζημιωθεί. Εάν όμως έρχεται ο άνθρωπος αυτός για δικό του λογαριασμό για να καταλάβει πώς δουλεύει, ε, για να καταλάβει καλύτερα πώς δουλεύει μια επιχείρηση, ε, εδώ είναι αυτονόητο ότι δεν χρειάζεται να αποζημιωθεί οικονομικά. υπάρχουν κάποια στάζ τα οποία διαρκούν λιγότερο από τρεις μήνες είναι στάζ για νέους και οι επιχειρήσει διαθέτει το χρόνο της για τη μαθητεία του νέου. Και υπάρχουν κάποια στάζ πάνω από τρει ε, μήνε που έχουν πιο επαγγελματικό χαρακτήρα και εδώ θα πρέπει βεβαίω να αμείβονται οι νέοι, να αποζημιώνονται. Και συμφωνώ ότι ορισμένε φορέ μερικοί εργοδότε παίρνουν ε, σταζιέρ, ανθρώπους που κάνουν στάζ, ε, μαθητευόμενους, για να αντικαταστήσουν τους κανονικά εργαζόμενους. Και εδώ θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Τώρα, ε, νομίζω ότι έτσι κι θα επανέλθουμε για τις συμβαστικέ τροπολογίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Τουρένεν. Είναι ουσιάδα στο θέμα, είναι καλή η έκθεση. Οι νέοι είναι το μέλλον μας και θα πρέπει να ασχοληθούμε μαζί τους, να εγγύψουμε στα προβλήματά τους. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Σέρκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ, όπως και η κυρία Μπρούνη, την έκθεση αυτή της κυρίας Τούρεν, η οποία μου φαίνεται εξαίρετη. Εγώ ε, κατέθεσα μία τροπολογία και μου έθεσε το σχετικό ερώτημα η κυρία Τουρέν γιατί κατέθεσα. Πρόκειται για το, την ε, τροπολογία παρθών 19, το F. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να θεωρήσετε ότι είναι ένα σχέδιο ε, συγγνώμη, ότι είναι ε, μια κοιλίδα σε μια ξεκάθαρη έκθεση αυτή η διατύπωση στην τελογική σκέψη F η οποία είναι εξαιρετικά συγκεχημένη το ελάχιστο και δεν είναι ένα θέμα των χωρών αλλά προκαλείται μία σύγχυση όσον αφορά τα ενεργά μέτρα προώθησης των νέων και τα παρουσιάζεται σαν παθητικά, μέτρα παθητικής φύσεως. Νομίζω ότι προκαλείται λοιπόν αυτή η σύγχυση και στην ε, ε, ισπανική διατύπωση λέει ότι είναι αυτά τα μέτρα η υπέτεια για το γεγονός ότι οι νέοι δεν μπορούν να έχουν μια ενήλικη και ανεξάρτητη ε, ζωής. Ε, ζωή. Εάν ε, τα πράγματα είχαν έτσι θα έπρεπε στη Δανία ή στη Μεγάλη Βρετανία τελικά να εξαλειφθούν αυτά τα μέτρα ούτως ώστε οι νέοι να έχουν μια ανεξάρτητη ζωή. Αυτό γράφει στα Ισπανικά. Ο τελόγος για τον οποίο οι νέοι δεν έχουν μια ενήλικη και ανεξάρτητη ζωή είναι ακριβώ αυτά τα μέτρα στήριξη των νέων. Εγώ νομίζω θα μπορούσαμε να κρίνουμε αυτά τα μέτρα ως επικίνδυνα από κάποιες μορφές που προσλαμβάνουν αλλά το να λέμε ότι δεν χρειάζεται να πάρουμε απολύτω κανένα μέτρο στήριξη παθητική ενεργητική ε, φύσεω, ε, στήριξη των νέων, θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο. Γιατί το συμπέρασμα που βγάζουμε από εδώ είναι ότι θα πρέπει να αφήσουμε ε, στην ελεύθερη αγορά το ζήτημα τη ένταξη των νέων σε αυτήν. Δεν ξέρω αν είναι το φταίξιμο τη μετάφραση στα ισπανικά, αλλά νομίζω ότι είναι μία παράγραφο αυτή που είναι γεμάτη από. προκαλεί σύγχυση και είναι εξαιρετικά επικίνδυνη είναι όσον αφορά τα περιθώρια ερμηνεία γιατί οδηγεί σε κάποιες λύσει αν όχι άκρα συντηρητικέ. Ε, ε, άκρο συντηρητικέ, συγγνώμη, αν όχι απλώς συντηρητικέ, άκρο συντηρητικέ. Ε, δεν ξέρω, ίσω είναι ένα θέμα φραστικής διατύπωσης. Ίσως είναι μόνο το πρόβλημα στα ισπανικά. Δεν ξέρω, είχαμε μια ακρόαση εδώ στην Επιτροπή και ήδη έγινε αυτή η επισήμανση ε, από τους νέους οι οποίοι δεν κατάλαβαν ε, ακριβώς τι σημαίνει και θεώρησαν ότι είναι επικίνδυνη. Grazie signora Presidente. Ho detto da Belline ringrazia il collega TI Rapporto. Ο κύριος Κάζα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ την ε, κυρία Τερεν για την εκθεσή τη. Εγώ έχω καταθέσει διάφορες τροπολογίες με στόχο να αποσαφηνίσω κάποιες θέσεις και επίσης να κάνω αυτό που λένε οι Άγγλοι προστιθέμενη αξία, value added. Δεν θα αναφερθώ σε κάθε μια τροπολογία χωριστά, αλλά θα ήθελα να μιλήσω εν γέννη για το τι προτείνω. Πιστεύω πως το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει και να επηρεάσει επίσης ιδιαίτερα όταν μιλάμε για ορόσημα για το μέλλον σε σχέση με την απασχόληση των νέων, σε σχέση δηλαδή με τη σύγκριση αποδόσεων. πριν να προσθέσουμε περαιτέρω χρήματα στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, θα πρέπει καταρχήν να δούμε μια ματιά, ε, να ρίξουμε μια ματιά και να δούμε πώς το Κοινωνικό Ταμείο θα γίνει πιο αποτελεσματικό, όχι απλά να αυξήσουμε την ε, οικονομική του στήριξη. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε το Ταμείο, να το κάνουμε πιο αποτελεσματικό. Πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους νέους να γίνουν πιο ανεξάρτητοι ιδιαίτερα όταν γίνουν ενήλικες. Και Βέβαια, εγώ δεν θεωρούμε πλέον νέος, αλλά έχω πολύ στενή επαφή με τους νέους και πιστεύω πως δεν είναι καθόλου εύκολο να αφήνει κανείς την σχολική του ζωή και να καταλήγει άνεργος. Η κυρία Γκρίνερ μίλησε για χαμηλά εισοδήματα, ε, για χαμηλούς μισθούς. Πώς ε, να φανταστεί κανείς το καθόλου μισθό. Τι εννοούμε τώρα όταν λέμε ενήλικη ζωή. Είναι κάτι το οποίο συζητήσαμε και στην προηγούμενη έκθεση και αφορά την χρήση της διαβίου κατάρτισης είναι πολύ κρίσιμο. Ωστόσο πρέπει να καταστεί πιο εύκολο για τους νέους. Όταν δηλαδή φεύγουν από το σχολείο, όταν τελειώνουν το σχολείο, να μην είναι αδύνατο να μπουν στην αγορά εργασία. Να ρίξουμε μια ματιά στις στατιστικές και να δούμε ότι ανάμεσα στην, σε όλους τους ανέργους που είναι πολλοί, οι νέοι είναι οι πρώτοι και δεν μειώνεται η ενεργεία στους νέους, αλλά αντίθετα αυξάνεται. Και αυτό που συμβαίνει σήμερα σημαίνει ότι αυτό που κάνουμε δεν επηρεάζουν τους νέους, δεν τους επηρεάζουν θετικά. Άρα αυτό πρέπει να σκεφτούμε. Τι πρέπει να κάνουμε, τι οφείλουμε να κάνουμε ώστε να βοηθήσουμε τους νέους. Να δούμε τι είδους αλλαγές μπορούμε να κάνουμε, πού θα βρούμε συμβαστικές λύσεις ώστε η ζωή των νέων να γίνει πιο εύκολη έτσι ώστε να συνδέσουμε την ε, διαδικασία της διαβίου κατάρτισης, να αναφέρω και την, ε, την τροπολογία της κυρίας Γκρούνη, την 37. Εγώ προσλέγω στο μέλλον με αισιοδοξία και ελπίζω πως μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα φτάσουμε σε κάποιες επιβαστικές λύσεις ώστε να είναι επιτυχής η έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η κυρία Ράπτη έχει το λόγο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, έχω την τιμή να είμαι σκιώδης εισηγήτρια από την πλευρά των σοσιαλιστών. Ε, θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω την Έμιλη για το πολύ καλό κείμενο που μας έδωσε. Διότι όταν κάποιος έχει ένα πολύ καλό κείμενο ως βάση, μπορεί να δουλέψει καλύτερα και μπορεί να δώσει τροπολογίες που να βελτιώνουν ακόμη περισσότερο το στόχο του κειμένου. Και ο στόχος του κειμένου, ο στόχος αυτής της έκθεσης είναι πάρα πολύ σημαντικός κατά τη γνώμη μου. Για τον πολύ απλό λόγο ότι η νέα γενιά είναι αυτή για την οποία εργαζόμαστε. Η νέα γενιά η σημερινή είναι μια ιδιαίτερη γενιά, ίσως είναι η πρώτη νέα γενιά που θα ζήσει δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξη, αλλά το τονίζω, ίσως είναι η πρώτη νέα γενιά που θα ζήσει χειρότερα από τους γονείς. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο κρίσης γενικότερης και οφείλουμε να τη λάβουμε υπόψη όταν συζητάμε για τους νέους και όταν σχεδιάζουμε για τους νέους έχοντας ρίξει μια ματιά στις τροπολογίες νομίζω και αισθάνομαι ότι υπάρχουν αρκετά περιθώρια πάρα πολλά περιθώρια θα έλεγα για συμβιβαστικές τροπολογίες. Ε, υπάρχουν μερικά σημεία που θέλουν διευκρίνηση θέλουν ε, κουβέντα και προβληματισμό όπως είναι ανάμεσα σε αυτά αυτό που ανέφερε ο συντονιστής μας των σοσιαλιστών ο κ. Σέρκας είναι ένα θέμα που πρέπει να μας προβληματίσει να δούμε πώς θα το χειριστούμε. Όπως από την άλλη μεριά υπάρχουν και προβλήματα ε, που πραγματικά νομίζω, όχι προβλήματα, να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη προβλήματα, υπάρχουν και κάποιες απόψεις που τουλάχιστον για τη δική μου, ε, από τη δική μου ματιά είναι προβληματικές. Αναφέρω ας πούμε ένα παράδειγμα, για να μην αναφερθώ σε όλες τις τροπολογίες, ένα, ένα ε, παράδειγμα είναι η τροπολογία 96. Μιλάω για την τροπολογία του κυρίου Χέλμερ που ζητά να βγει ένα, μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση από την παράγραφο 11. Είναι η πρόταση που λέει «Υπογραμμίζει ότι η ευελιξία χωρίς κοινωνική ασφάλεια δεν αποτελεί αηφόρο τρόπο καταπολέμησης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην αγορά εργασίας. Αυτό το κείμενο, αυτό το κομμάτι, ο κύριος Χέλμαρ ζητάει να διαγραφεί. Κατά τη δική μου γνώμη είναι ε, κεντρική ιδέα που πρέπει να παραμείνει στο κείμενο, γιατί αν βγάλουμε αυτό το κομμάτι μέσα από την παράγραφο 11, είναι πραγματικά σαν να αφήνουμε τη νέα γενιά ανυπεράσπιστη στο έλεος των εργοδοτών. Ε, το αναφέρω σαν ένα παράδειγμα που χρειάζεται πολύ πολύ μεγάλη προσοχή στον τρόπο που θα το χειριστούμε. Απ' την άλλη πλευρά βλέπω με χαρά ε, τροπολογίες ε, από όλες τις πολιτικές ε, ομάδες που α, ε, κατατείνουν στο να μπορέσουμε να κάνουμε πιο εύκολη την είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας και βέβαια δεν μπορώ να μην μπω στον πειρασμό ε, να πω πόση σχέση έχει η έκθεση αυτή που ετοιμάζουμε τώρα με την έκθεση που συζητήθηκε προηγουμένως σε σχέση με τις άτυπες μορφές εργασίας, με τις άτυπες συμβάσεις. Και αυτό γιατί. Διότι συνήθως στις άτυπες συμβάσεις αυτοί οι οποίοι είναι τα θύματα, χρησιμοποιώ τη λέξη θύματα εντός εισαγωγικών, είναι οι νέοι είναι οι νέοι οι οποίοι προσπαθώντας να ανοίξουν μια χαραμάδα, μια πόρτα για να μπουν στην αγορά εργασίας, πάρα πολλές φορές δέχονται να καταπατώνται δικαιώματά τους, δέχονται ε, διάφορες διακρίσεις και διάφορες υποχρεώσεις και πιέσεις από την πλευρά των εργοδοτών. Αυτά όλα πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας. Ε, για να κλείσω και να είμαι ε, σύντομη, ε, αισθάνομαι αισιόδοξη για την πορεία αυτής της έκθεσης. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να προωθήσουμε ακόμη περισσότερο το κείμενο που έχει φτιάξει η Έμιλη και να καταλήξουμε ε, σε ένα κείμενο που πραγματικά θα μπορέσει να δεσμεύσει θετικά για τους νέους την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ. Ähm, ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στην εισηγήτρια για να απαντήσει σε αυτά που ακούστηκαν. Εντάξει. Ευχαριστώ. Σύντομα, σας ευχαριστώ για όλες τις παρατηρήσεις που έγιναν. Τις σημειώνω. Πολύ σύντομα θα συναντηθούμε σε συνάντηση των σχεδόντων εισηγητών. Θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτό που είπε η κυρία Ράπτη για την 96, ε, την ασφάλεια. Χρειαζόμαστε την πρόταση αυτή και πιστεύω ότι θα βρει την υποστήριξη της Επιτροπής. Και μια τελευταία παρατήρηση πάλι για το εκτιμώντας σίγμα ταφ. Ποτέ δεν με κατηγόρησαν στο παρελθόν ότι είμαι συντηρητική. Πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό. Αλλά ναι, μου συνέβη και αυτό. Να σας ευχαριστήσω κύριε Τσέρκας. Εγώ το πρόβλημα που βλέπω στα τρία αυτά παραδείγματα είναι ότι οι νέοι έχουν λιγότερη προστασία, επειδή είναι νέοι, από ότι άλλοι εργαζόμενοι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στη Δανία έγινε μεταρρύθμιση περίπου πριν 10 χρόνια, που σήμαινε ότι αν κάποιος ήταν κάτω των 25 ετών, ε, δικαιούτο μόνο το 50% του κανονικού επιδόματος ανεργίας. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος είναι νέος χτίστης, έχει λάβει επαγγελματική κατάρτιση, μπορεί να δουλεύει επί δύο χρόνια. Γίνεται η παγκόσμια κρίση, η οικονομική κρίση όπως η παρούσα και πηγαίνει κανείς στο κέντρο εργασίας και λέει ότι αν δεν έχω δουλειά, λαμβάνει μόνο το 50% του επιδόματος ανεργία. Γιατί, επειδή είναι κάτω των 25 ετών. Αυτό το θέμα θέλω να θίξω. Το ίδιο ισχύει για τον κατώτατο μισθό στο Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι πολύ χαμηλός και είναι πραγματικά, νέο για τους, είναι πραγματικά πρόβλημα για τους νέους να ε, βγάλουν αρκετά λεφτά. Να έχουμε διαφορετικό κατώτατο μισθό για τα άτομα κάτω των 25 ετών ή να έχουμε έναν εθνικό βασικό μισθό. Τελευταίο παράδειγμα, στη Γαλλία. Και μπορεί να χρειαστεί να το συζητήσουμε αυτό κάπως. Καταλαβαίνω ότι αυτό συμβαίνει επειδή θέλετε να σπρώξετε τους νέους στην ε, απασχόληση, ε, να τους εντάξετε στην κοινωνία. Το, η ίδια ιδέα υπήρχε στην Δανία, αλλά σε στην οικονομική κρίση μπορεί να έχει ολοκληρώσει κανεί τι σπουδέ του, να είναι κάτω των 25 ετών και στην ε, Δανία να δικαιούται πάρα πολύ λίγα ή πολύ λίγα στη Γαλλία. Και για μένα αυτό είναι πρόβλημα. Ή, ή για τίποτα στη Γαλλία. Διότι μπορεί κανεί να ψηφίσει, έχει τι ίδιε υποχρεώσει, ε, πληρώνει φόρου. Έχει λοιπόν κανεί τι ίδιε υποχρεώσει, όχι όμω τα ίδια δικαιώματα. σω θα πρέπει να εξετάσουμε την διατύπωσε. Είμαι διατεθειμένη να το κάνω αυτό. Δεν νομίζω ότι όμω θα πρέπει να φοβηθούμε να αναφέρουμε τα παραδείγματα των περιπτώσεων όπου υπάρχουν προβλήματα. Πιστεύω όμω ότι μπορούμε να βρούμε μια λύση. Αυτή ήταν η τελευταία παρατήρηση. Όχι, μία ακόμα παρατήρηση. Γνώρισα έναν νεοχτίστη στη Δανία. Αυτό ήταν το παράδειγμα που σα ανέφερα πριν. Ζούσε σε μια μικρή πόλη που λέγεται Σλέελ στη Δανία. Δεν έχει δουλειά, διότι δεν υπάρχει δουλειά καθόλου για χτίστε, για οικοδόμου στη Δανία. Ε, σχεδόν το 50% των ε, χτιστών ε, είναι άνεργοι. Πριν κάποια χρόνια αγόρασε ένα ε, διαμέρισμα με την κοπέλα του. Έχουν ανεξάρτητη ζωή ως ενήλικες, ε, αλλά τώρα ε, λαμβάνει μόνο το 50% του επιδόματο ενέργεια και οι γονεί του πληρώνουν το ε, διαμέρισμα, επειδή αλλιώ θα πρέπει να το φύγει. Και δεν είναι κανένα τεράστιο διαμέρισμα, είναι ένα μικρό διάρρη σε μια μικρή πόλη στη Δανία. Αυτό είναι που θέλω να σας πω. Αυτό εννοώ όταν λέω ότι δεν μπορεί κανείς να ζήσει ανεξάρτητα ως ενήλικας. Ευχαριστώ και προσβλέπω στην καλή συζήτηση. Ωραία. Έτσι ολοκληρώσαμε αυτή τη συζήτηση και θα ψηφίσουμε στις 31. Όχι. Α. Ωραία, κοιτάω τώρα το σωστό πίνακα. 1η Ιουνίου θα έχουμε πάλι το θέμα στην ημερήσια διάταξη, θα συζητηθούν οι συμβαστικέ προπολογίες και την επόμενη μέρα, 2 Ιουνίου δηλαδή, θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή και προβλέπεται για την Ολομέλεια του Ιουλίου η έκθεση αυτή. Ολοκληρώσαμε έτσι τη συζήτηση. Και τώρα φτάνουμε σε μια πολύ δύσκολη περίπτωση, διότι θα πρέπει ε, να παρουσιάσω τη δική μου έκθεση ε, και να προεδρεύω ταυτόχρονα. Λένε ότι οι γυναίκες μπορούν να τα κάνουν αυτά, διότι είναι πολύ καλές στο multitasking. Αυτό θα κάνω λοιπόν. Θα μου δώσω λοιπόν το λόγο. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομη και πιο συγκεκριμένη, ώστε να δώσω τη δυνατότητα στους παρόντες να συζητήσουν την έκθεση. Πρόκειται πάλι για έκθεση πρωτοβουλίας. Τίτλο έχει την ανάπτυξη του δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας νέας βιώσιμης οικονομίας. Το πρώτο που σκέφτηκα ε, τι περιμένουμε από την έκθεση αυτή. Ε, στοιχεία σχετικά με το πόσες επασχόλησεις έχουν δημιουργηθεί στον ε, κάθε τομέα. Κατέβαλα προσπάθειες να βρω τα σχετικά στοιχεία, να τα αξιολογήσω αντικειμενικά και ήθελα να τα συμπεριλάβω στην έκθεση. Αλλά η αξιολόγηση έδειξε ότι υπάρχουν πολλές προϋποθέσεις ε, σχετικά με τα νούμερα αυτά. Μιλάμε δηλαδή καταρχήν ποιο είναι ο των θέσεων, ε, των θέσεων απασχόλησης, ποια νούμερα ισχύουν μετά τη μελέτη περίπου 20 ερευνών κατέληξα ότι Είναι δύσκολο να παρουσιάσω τα νούμερα και παρουσιάζω την όλη διαδικασία στην έκθεση. Το θέμα είναι δηλαδή πώς ορίζουμε τη θέση απασχόλησης. Προσπαθήσαμε να καταλήξουμε σε έναν ορισμό Καταλήξαμε σε έναν ορισμό που πιστεύω ότι θα βρει τη συμφωνία όλων και προέρχεται από το διεθνές έγγραφο του ILO τη Διεθνούς Οργάνωση Εργασία και προτάθηκε για τους Υπουργού Εργασία των G8. Νομίζω ότι ο ορισμός αυτός είναι διεθνώς αναγνωρισμένος και μπορούμε να τον υιοθετήσουμε. Ο ορισμό αυτό, λέει ότι κάθε θέση απασχόληση είναι πράσινη εφόσον συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος στην μείωση κατανάλωσης ε, και στη, στο πιο καθαρό αέρα και στο πιο καθαρό περιβάλλον. Μπορεί δηλαδή να είναι μια θέση απασχόληση σε μια διαδικασία παραγωγής. μέσω της οποίας να φτάνει άλλο προϊόν σε μας. Είναι λοιπόν ανοιχτός και ευρύς ο ορισμός αυτός είναι λοιπόν σαφές ότι μιλάμε για ε, νέες θέσεις απασχόλησης αλλά και για θέσεις απασχόλησης παλιές οι οποίες όμως έχουν βελτιωθεί. Έτσι λοιπόν η οπτική μας είναι κάπως διαφορετική και θα προτιμούσα ακριβώς αυτή την οπτική. Η δεύτερη πτυχή που εξετάζω είναι το γεγονός ότι οι νέοι τομείς εμφανίζονται σαν μανιτάρια και είναι τελείως ξεκομμένοι από αυτό που ονομάζουμε εμείς τον εργασιακό κόσμο της ε, ε, Ευρώπης. Ε, κάπου δηλαδή όπου πραγματοποιείται εργασιακός διάλογος, κοινωνικός διάλογος και που υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκε εργασίας. Οι κοινωνικοί εταίροι αγνοούν τις νέες αυτές θέσεις απασχόλησης, δεν έχουν προσέξει καν ότι εμφανίζονται τέτοια φαινόμενα. Δεν έχουν δημιουργηθεί λοιπόν οι απαραίτητε συνθήκες πλαίσιο. Γι' αυτό απευθυνόμαστε στους κοινωνικού εταίρους. Το αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της γρήγορης εμφάνισης αυτών των φαινομένων είναι ότι υπάρχουν προβλήματα στους συγκεκριμένους τομείς. Δεν πιστεύω ότι αυτό δίνει καλή εικόνα των νέων τομέων, των ε, πράσινων τομέων, εάν ισχύει το δίκαιο του, της Άγριας Δύσης. Θα πρέπει οι θέσεις αυτές που δημιουργούνται να είναι θέσεις από τις οποίες να μπορεί να ζήσει κανείς και να είναι βιώσιμες. Και γι' αυτό έχω συνδέσει αυτά τα δύο πράγματα μεταξύ τους. Και γι' αυτό έχω αναθέσει κάποια καθήκοντα στους κοινωνικούς εταίρους. Πρόκειται για μια συζήτηση την οποία ήδη έχουμε κάνει υπό διάφορες μορφές, είναι πολύ ενδιαφέρουσα και ε, πιστεύω ότι μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε στην συζήτηση αυτή. Άλλο ε, σημείο σημαντικό είναι ένα έγγραφο για το θέμα αυτό ένα έγγραφο τη Επιτροπής που ονομάζεται Απασχόληση 2009 το οποίο περιλαμβάνει ολόκληρο κεφάλαιο σχετικά με την αλλαγή του κλίματος σε σχέση με, τις, με την απασχόληση, κλιματική αλλαγή και απασχόληση. Αλλά αυτά που υπάρχουν στο έγγραφο αυτό παραμείναν θεωρία. Και η Ευρώπη έχει μάθει πολύ λίγα τελικά από τις ε, σχετικές εμπειρίες. Το έγγραφο της Κομισιόν έχει δημιουργήσει μόνο θεωρητικές εικόνες και όχι πραγματικές. Ένα παράδειγμα είναι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπου υπάρχουν στοιχεία τα οποία βασίζονται στην θεωρητική κατάσταση όταν ε, χάνεται μία θέση ε, απασχόλησης ε, με μεγάλες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα πόσα άλλες δημιουργούνται στη θέση της. Αυτό δεν βασίζεται σε πραγματικούς ανθρώπους. Ε, υπάρχουν ε, εμπειρίες σχετικά με τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Ε, στην Γερμανία προωθείται η ανανεώσιμη ενέργεια και οι θέσεις που δημιουργούνται είναι περισσότερες από όσο διαπιστώνει η Κομισιόν. Είναι λοιπόν πολύ ενδιαφέρουσα η εξέλιξη. Θα το δείτε αυτό. Πολύ ευχαρίστω θα δώσω το έγγραφο αυτό στους σκιώδεις συζητητές και στους συναδέλφους, διότι οι εξέλιξεις δείχνουν ότι Υπάρχει μια τεράστια εξαγωγική αγορά η οποία δημιουργεί πολλές περισσότερες θέσεις εργασίας από αυτές που χάνονται. στην εξαγωγή ε, ε, πράσινης ενέργειας η Ευρώπη είναι ανταγωνιστική. Θα πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη μας. Το τελευταίο θέμα και το σημαντικότερο για μένα είναι πώς θα φτάσουμε μέχρι εκεί να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε αυτό το ε, δυναμικό. Δύο ε, πράγματα. Πρώτον, χρειαζόμαστε σταθερέ συνθήκε πλαίσιο, διότι ε, έχει αποδειχθεί ότι στι χώρε όπου υπάρχουν αυτέ οι σταθερέ συνθήκε πλαίσιο και μάλλον στις χώρες και στους τομείς όπου δεν υπάρχουν αυτές οι σταθερές συνθήκες πλαίσιο δεν ε, γίνεται εκμετάλλευση του δυναμικού. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση και γι' αυτό έχω συνομιλήσει με ε, τις άλλες επιτροπές που είναι υπεύθυνες, για, που είναι αρμόδιες για τον τομέα αυτό και ε, τους έχω ζητήσει να εξετάσουν την ε, γνωμοδότηση. Το τελευταίο θέμα είναι το θέμα του ειδικευμένου ε, εργατικού δυναμικού που έχει να κάνει με την ε, μη ε, εκμετάλλευση των αποθυμάτων τον, του δυναμικού. Βλέπετε εδώ πέρα έναν πίνακα που δείχνει εντυπωσιακή εξέλιξη. Γιατί δεν έχουμε ειδικευμένο προσωπικό, επειδή δεν δίδεται αρκετή προσοχή στο θέμα της εκπαίδευσης. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε πώς μπορούμε να πετύχουμε στους νέους τομείς αλλά και στους τομείς όπου γίνονται τροποποίησεις ε, στις θέσεις ε, απασχόλησης για να ε, πετύχουμε την πράσινη οικονομία πώς μπορούμε να έχουμε συνεχή μετεκπαίδευση και πώς μπορούμε να ε, τους μεταδώσουμε αυτό το αίσθημα της ευθύνης για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε το δυναμικό. Αυτά είναι τα βασικά σημεία της έκθεσης. Ε, περιμένω τώρα να ακούσω τη συμβολή των, ε, της παρεμβάσης των ε, συναδέλφων. Ε, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που παρέμειναν παρότι είπαν ότι δεν είχαν αρκετό χρόνο. Έχω ήδη κάποιον στον κατάλογο των ομιλητών. Ο κύριος Λούντβιξον, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω ε, και την ε, εισηγήτρια. Ένας λόγος που παρέμεινα είναι ότι θα προλάβω να επιστρέψω στο Γκέτεμπορκ παρά ε, την παραμονή μου. Όπως ξέρετε δεν συζήτιεται πια το ότι είναι σημαντικό να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε, τον τρόπο που παράγουμε και καταναλώνουμε προϊόντα. Η πράσινη οικονομία είναι ένας σαφής στόχος, τον οποίο δεν μπορούμε να αποφύγουμε αν θέλουμε να μειώσουμε την αλλαγή του, ε, τις επιπτώσεις αλλαγής του κλίματος. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν συζητάμε αν θα πρέπει να το κάνουμε, αλλά πώς θα το κάνουμε και πώς θα πετύχουμε τις ε, σημαντικές αυτές αλλαγές. Σχεδόν καθ' όλη την επαγγελματική μου, ε, σχεδόν καθ' την ε, επαγγελματική μου σταδιοδρομία εργάστηκα στον τομέα των οχημάτων και παρακολουθώ την προσπάθεια με, ε, μετατροπής στην πράσινη οικονομία. Σημαντικό είναι η πράσινη οικονομία να έχει μακροπρόθεσμους και σαφείς κανόνες ώστε να υπάρχουν σαφή κίνητρα για να αλλάξει ο τρόπος παραγωγής. Θα πρέπει να μπορούμε να υπολογίσουμε το κόστος να προσαρμοστούμε στο μέλλον. Οι τροποποιήσει θα πρέπει να γίνουν γρήγορα για να πετύχουμε καλό αποτέλεσμα, αλλά και σε ρυθμό, ώστε η βιομηχανία να έχει το χρόνο να σχεδιάσει το μέλλον και να ε, αναδιαρθρωθεί. Η γρήγορη αλλαγή θα ε, συνεπάγεται και καλύτερα νούμερα τελικά στον ισολογισμό και αυτό είναι καλό. Αλλά Υπάρχουν και βιομηχανίες που έχουν μακρύτερο χρονικό διάστημα προγραμματισμού και θα πρέπει να υπάρχει κάποια ευελιξία. Άλλο σημαντικό θέμα στην προσαρμογή στις ε, πράσινες θέσεις εργασίας ε, είναι να εξετάσουμε το συνολικό του κύκλου ζωής του προϊόντος. Και δεν θα πρέπει μόνο η διαδικασία παραγωγής να γίνεται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Το ίδιο το, περιβάλλον θα πρέπει να, το, το, ίδιο το προϊόν θα πρέπει να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Θα πρέπει να παράγεται με τρόπο ώστε να μπορεί να ανακυκλωθεί με λογικό τρόπο. Και ο χειρισμός του επίσης να είναι φιλικός προς το περιβάλλον. Συμφωνώ με την εισηγήτρια σχετικά με τη σημασία των αξιοπρεπών θέσεων εργασίας στους νέους τομείς. Πολύ συχνά μιλάμε για πράσινες ε, θέσεις απασχόλησης και αναφερόμαστε σε θέσεις ε, εργασίας ε, υψηλή τεχνολογία. Υπάρχουν όμως και θέσεις απασχόλησης χαμηλότερης εξειδικευσής. Σημαντικό είναι ότι όταν μιλάμε για νέους τομείς ε, μπορεί να μιλάμε για τομείς ε, με χαμηλές απαιτήσεις ως προς, τον, ε, προς την διοργάνωση. Θα χρειαστούν προσπάθειες ως προς την κατάρτιση για να μπορέσει να γίνει το πέρασμα προς τις προς τις πράσινες θέσεις Επίσης θα χρειαστεί τεχνολογία εχμής καθώς και περισσότερη κατάρτιση. χρειάζεται προσαρμογή των δεξιοτήτων που ήδη υπάρχουν. Δεν χρειάζεται να δημιουργηθούν νέε δεξιότητε. Πιστεύω ότι η έκθεση αυτή είναι ε, καλή βάση για τη συνέχιση των ε, συζητήσεων και περιμένω να ακούσω τι ε, απόψει των συναδέλφων. Δυστυχώ θα πρέπει να φύγω. Οι παρεμβάσει όμω θα σημειωθούν και θα τι εξετάσω εκ των υστέρων. Σα ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ που αντέξατε τόσο πολύ και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Äh, Συνάδελφο Ζάι, θα ήθελα να σας δώσω το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, Συσυχητρία. γιατί μπορέσαμε όντω να συνεδριάσουμε και να ενημερωθούμε εκ των προτέρων όσον αφορά τις λεπτομέρειες του θέματος. Γιατί η έκθεση αυτή είναι πολύ σοβαρή και πρέπει να μπορούμε να μιλήσουμε και να ορίσουμε με κοινό τρόπο τι είναι μια βιώσιμη θέση, μια πράσινη θέση απασχόλησης και ούτω καθεξής. Εγώ προσωπικά μιλώ περισσότερο για μια απασχόληση σε μια βιώσιμη οικονομία, γιατί μια πράσινη ε, θέση ήδη χρησιμοποιείται από κάποια άλλη ομάδα στο Κοινοβούλιο. Να υπογραμμίσω εδώ, ανάμεσα στα όσα υπογράμμισε και η συγγύτη, ότι είναι πολύ δύσκολο να ορίσουμε μια θέση, μια άλλη ή κάποιο συγκεκριμένο τομέα που θα μπορούσε να είναι πιο πράσινος από άλλους και να αποκλείσουμε κάποιους άλλους τομείς. Γι' αυτό και πιστεύω πως είναι εξαιρετικά σημαντικό να μπορέσουμε να έχουμε μια προσέγγιση πολύ πιο ευρεία από αυτή που προτείνει η εισηγήτρια. Στην ε, παραδοσιακή τώρα βιομηχανία, ας πούμε για την ε, αυτοκινητοβιομηχανία, ε, για την κατασκευή ελαστικών, θα μπορούσαμε και να πούμε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται λιγότερες πρωτεσίλες, 10% λιγότερο ή 20% λιγότερο, αυτά σε έναν τομέα παραδοσιακό, όπου μπορούμε όμως να υιοθετήσουμε βιώσιμες λύσεις. Όμως τι πρόβλημα προκύπτει στις στατιστικές, ιδιαίτερα για την αριθμητική μέτρηση μιας βιώσιμης θηγατρικής, υπάρχει πρόβλημα και εσείς οι ίδιοι το αναφέρατε. Επίσης αυτό που είπατε είναι ότι όταν υποστηρίζεται ένα τομέας μπορεί να υπάρξει στρέβλωση. Ορισμένοι δηλαδή υποστηρίζουν, άλλοι όχι. Ε, υπάρχουν φορολογικά κίνητρα ας πούμε τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επενδύσεις κακής ποιότητας, δηλαδή αρνητικές. Δηλαδή μπορεί να στηρίξουμε ένα τομέα μόνο ο τομέας αυτός συνηθίζει στην στήριξη κατά κάποιο τρόπο και τελικά θέλει να συνεχιστεί. Όταν όμως η στήριξη σταματήσει, ο τομέας καταραίει. Θα πρέπει να υπάρξουν λοιπόν κάποιες ε, προσαρμογές και θα πρέπει να μιλήσουμε για τέτοιου είδους καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν. Στη συνέχεια θα ήθελα κάπως να επικρίνω την προσέγγιση της ηγήτριας όσον αφορά το θέμα της ποιότητας αυτών των θέσεων απασχόλησης. διότι μιλάμε για κακοπληρωμένες ε, θέσεις. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις συνθήκες εργασίας αυτών των εργαζόμενων Πρέπει δηλαδή πραγματικά να λάβουμε υπόψη τι ηθίκε εργασία και να αποφύγουμε το dumping. Και σίγουρα θα πρέπει να γίνει dumping όσον αφορά την ποιότητα των συμβάσεων εργασία. Και αυτό σε όλα τα κράτη-μέλη. Σε όλα τα κράτη-μέλη οι συλλογικέ διαπραγματεύσει στόχο έχουν να πλαισιώσουν αυτέ ε, τι θέσει απασχόληση, αυτέ τι βιώσιμε θέσει ή πράσινε θέσει να ληφθούν υπόψη και να εξεταστούν με τον ίδιο ακριβώ τρόπο όπω και οι υπόλοιπε θέσει. Και επίσης έχω την εξή ερώτηση. Η συγκίτρια ελαφρώς επέκανε το γεγονός ότι θα πρέπει να φτάσουμε στο 40% του πληθυσμού ή των νέων με ένα δίπλωμα ανώτατης εκπαίδευσης, ένα πανεπιστημιακό δίπλωμα, μα 40% ε, είναι ένα στόχο στον οποίο θα πρέπει να επιτύχουμε, αλλά Σίγουρα θα πρέπει να υπερκαταρτίζουμε τους πολίτες μας, αλλά να έχουμε πάντα υπόψη το γεγονός ότι όλο ένα και περισσότεροι νέοι πρέπει να καταρτίζονται, να εκπαιδεύονται και να ε, παρακολουθούν κατάρτιση καθόλου τον επαγγελματικό του βίο. Εγώ προέρχομαι από τη Σκανδιναβία. Είμαι συνηθισμένη στο γεγονός ότι στην πολιτική της ισότητας στις ε, σκανδιναβικές χώρες έχουμε προχωρήσει πολύ και ότι οι γυναίκες εργάζονται περισσότερο στις βόρειες χώρες και αυτό το καταφέραμε χωρίς ποσοστώσεις. Από τους Φινλανδούς ε, βουλευτές οι περισσότεροι Περισσότερες είναι γυναίκες, δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με ποσοστώσεις. Ε, νομίζω πως θα πρέπει να καταθέσω μια σχετική τροπολογία. Τρίτο στοιχείο ελαφρώς επικριτικό αφορά το θέμα του ότι αναφέρεται τον φόρο το BIN. Με ποιο τρόπο Δηλαδή μπορεί κανεί να συλλέξει ε, κονδύλια. Εγώ μέσα στην κρίση που διανύουμε είμαι κατά μια τέτοια ιδέα. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε νέου φόρους που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε στρέβλωση της αγοράς εργασίας. Η δημόσια οικονομία στα κράτη-μέλη πρέπει να αντιμετωπίσει τεράστιες προκλήσεις. Δεν νομίζω πως υπάρχει λόγος λοιπόν για να υποστηρίξουμε κάτι τέτοιο και έπειτα όταν Μιλάμε για νέο τομεί της βιώσιμης, της βιώσιμης οικονομίας, το οποίο ορισμός είναι κάπως αόριστος. Ενώ επενδύουμε σε αυτόν πολλές ελπίδες, το σημαντικό είναι να θυμάται κανείς ότι Στην πρώτη παράγραφο της έκθεσης λέμε ότι είναι οι λειτουργίες, ο τρόπο παραγωγής του κάθε τομέα που καθορίζουν κατά πόσο αυτός ο τομέας, ο κλάδος είναι βιώσιμος ή όχι. Το να επενδύσουμε λοιπόν σε νέους ε, βιώσιμους ε, κλάδους που δεν είναι κατάλληλα καθορισμένοι είναι οριστό και γενικό. Φαντάζομαι πω θα λάβουμε διάφορε τροπολογίε που θα βελτιώσουν την έκθεση και ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια γιατί η έκθεσή τη πραγματικά ε, προκάλεσε την προσοχή μα. Ευχαριστούμε πολύ κυρία συνάδελφε. Ο κύριο Ένιελ έχει το λόγο. Ναι, στην ίδια την έκθεση θα ήθελα να πω το εξή Είναι πετυχημένη και μια εξαιρετική βάση για την περαιτέρω εργασία. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι το οποίο είπε η κυρία Σρέτερ κάποτε προφορικά. Επικρίνει το γεγονός ότι οι κοινωνικοί εταίροι δεν έχουν ασχοληθεί με τις νέες μορφές βιομηχανίας. Δεν τις έχουν καν λάβει υπόψη τους. Ε, αυτό θέλω να αμφισβητήσω, αλλά νομίζω ότι είναι μόνο ένα τμήμα της αλήθειας. Ε, στη βάση της μου εμπειρίας στην αιωλική ενέργεια όχι μόνο εκεί, αλλά και σε άλλες νέες επιχειρήσεις πολύ συχνά η τήρηση των κοινωνικών ε, προδιαγραφών η εκπροσώπηση των εργαζομένων μέσω εργασιακών συμβουλίων θεωρούνται ως κολλήματα σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις και πολλές φορές ε, εμποδίζουν τους εργαζόμενους να σαν εκπροσωπηθούν μέσω των συνδικάτων ή των επιχειρησιακών συμβουλίων. Έχω την εντύπωση ότι στο κεφάλαιο ε, δίκαιη κοινωνική αλλαγή ε, όταν ε, αφορά την ανάθεση έργου σε τέτοιου είδου επιχειρήσεις να εξετάζει κανείς κατά πόσο τηρούνται τέτοιου είδου κοινωνικές προδιαγραφές ως κριτήρια για την ανάθεση έργου. Ε, νομίζω ότι στην ε, πιο παραπέρα συζήτηση αυτής της έκθεσης ίσως ε, καταλήξουμε σε μια πιο ενδεδειγμένη διατύπωση που να περιλαμβάνει ακριβώς αυτή την πτυχή. Ε, δεν ξέρω. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Η Επιτροπή έχει τώρα το λόγο. Δεν ξέρω. Βρίσκεται εδώ ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής. Όχι. Και όμως κάποιος είναι εδώ. Η Μόνικα Σλέμπιγκερ. Δίνω στην Επιτροπή λοιπόν στο λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και συγγήτρια. Θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω για αυτή την ε, καλά δομημένη έκθεση. Η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης από την οποία προέρχομαι χαιρετίζει αυτή την πρωτοβουλία και συμμερίζεται πολλές ανησυχίες που εκφράζει η έκθεση, ειδικά όσον αφορά τις πιο ευάλωτες ομάδες ε, της αγοράς ε, εργασίας που θα πρέπει να μπορούν να υποφεληθούν από τις ε, περιβαλλοντικές προκλήσεις. Νομίζω ότι πολλά από τα αιτήματα που θέτει η έκθεση είναι θεμητά. Παρ' όλα αυτά θα το εκτιμούσαμε αν η έκθεση θα έχει αναγνώριση ορισμένε πρωτοβουλίε τη Κομισιόν, ιδιαίτερα όσον αφορά την πολιτική, ε, την χάραξη μια πολιτική απασχόληση που είναι σημαντική όσον αφορά την προσαρμογή στις νέες συνθήκες αγοράς εργασίας και οικονομίας. Θα ήθελα στην παρουσίασή μου να εστιάσω ε, σε κάποια σημεία, αλλά θα μπορούσα να σας διαβάσω και γραπτά αν το επιθυμείτε. Ε, καταρχήν, η στρατηγική Ευρώπη 2020. Η βιώσιμη μεγέθυνση, είναι ε, μία από τις τρεις ε, σημαντικές προτεραιότητες και η βιώσιμη ανάπτυξη δεν αφορά μόνο μία καλύτερη εξοπλίση των πόρων και πράσινη οικονομία, αλλά και μία ανταγωνιστική οικονομία, δηλαδή μία οικονομία που να υποστηρίζει και να ενισχύει τη θέση της Ευρώπης μέσω της ε, δημιουργίας και νέων αγορών. Ε, βεβαίως υπάρχει και άλλη προτεραιότητα ε, που είναι μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, δηλαδή που να διασφαλίζει πρόσβαση και ευκαιρίες για όλους στη διάρκεια του κύκλου ζωής τους και με τον τρόπο αυτό υποστηρίζοντας και διαχειριζόμενοι την αλλαγή. Στην ατζέντα για νέες δεξιότητες στοχεύει ακριβώς την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, ούτως ώστε να προσπαθούν καλύτερα οι εργαζόμενοι στις νέες συνθήκες και μεταξύ των προτεραιοτήτων της νέας στρατηγικής επελαμβάνεται και αυτή η προτεραιότητα η οποία αναφέρεται και στις ε, νέες κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν την απασχόληση και την οικονομία. Το θέμα των ε, δεξιοτήτων το αντιμετωπίζουμε ως εξής. Πιστεύουμε ότι η πρωτοβουλία για τις νέες δεξιότητες έχει οδηγήσει σε σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά τις μελλοντικές ανάγκες, ε, ε, τη μελλοντική ανάγκη της αγοράς ε, για νέες πράσινες δεξιότητες και μια επιτυχημένη και αποτελεσματική προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος. Για παράδειγμα, έχουμε κάποια προγράμματα για νέες δεξιότητες μέχρι το 2020. Ε, το πρόγραμμα ΕΣΚΟ έχει ήδη εκπονηθεί ε, που αφορά ένα ε, λεξικό το οποίο συνδέει τις νέες δεξιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση. Σε σχέση με τις νέες δεξιότητες θα ήθελα να πω οι τελευταίες προβλέψεις του ΣΕΝΤΕΦΟΠ λένε ότι θα υπάρξει αυξανόμενη ζήτηση ε, στα άνω, ε, στις ανώτερες και κατώτερες θέσεις εργασίας και μια στασιμότητα στις μεσαίες θέσεις εργασίας. Τώρα, τι σημαίνει αυτό για τις εξότητες όσον αφορά τις πράσινες θέσεις απασχόλησης. Βεβαίως, εδώ όλες οι δεξιότητες θα είναι αναγκαίες και οι ψηλές και οι χαμηλές, χαμηλού επίπεδου. Αλλά όσο αφορά τα περιβαλλοντικά προγράμματα, μία μελέτη της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας ε, Συνδικάτων έδειξαν ότι οι περιβαλλοντικές πολιτικές στην, στην αρχική τους φάση προκαλούν ε, ζήτηση για πιο υψηλές δεξιότητες γιατί υπάρχει ανάγκη νέων ε, τεχνικών και τεχνολογιών που θα εφαρμοστούν και ζήτηση για καινοτομίε. Βεβαίω, όταν θα ρημάσουν αυτέ οι δεξιότητε, θα υπάρξει χώρος και για τις χαμηλότερου επίπεδου δεξιότητες και για τις μεσαίες, ε, μεσαίου επίπεδου δεξιότητες υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει επαρκής κατάρτιση και εκπαίδευση. Και θα ήθελα εδώ να κλείσω την ε, συμβολή μου στη συζήτηση αυτή δίδοντας ορισμένες επιπρόσθετες πληροφορίες για την έκθεση για την απασχόληση την, ε, στην Ευρώπη το 2009 που προσπαθεί να δώσει μια υποπτία των διαφόρων μελετών ε, δηλαδή κυρίως για μια πιο αναλυτική προσέγγιση ερευνών της Επιτροπής αλλά και άλλων οργανισμών που αξιολογούν ε, τις επιπτώσεις της απασχόλησης στις κλιματικές ε, μεταβολές. Η σύγκριση με τα δικά σας συμπεράσματα δείχνει ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνουν ε, ξεκάθαρα ε, να διατυπώνουν ξεκάθαρα συμπεράσματα όσον αφορά αυτέ τι μεταβολέ. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει σύγκριση μεταξύ των διαφόρων μελετών, γιατί ακολουθούν διάφορε μεθοδολογικές προσεγγίσει, αναφέρονται στι διαφορετικέ ε, γεωγραφικέ περιοχέ κλπ. Παρόλα αυτά, θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή μου σε ένα καλό πιστεύω παράδειγμα μιας έρευνας η οποία αναλύει ειδικά την ευαισθησία των εξαγωγών και της ε, ε, ε, μια έρευνα που έγινε το 2009 από το Verhoeven Ινστιτούτο και οι οποίοι παρουσιάζουν διάφορα σενάρια των, του μεριδίου, του, της μελλοντικής κατανομής των μεριδίων στην ευρωπαϊκή αγορά όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έχουν ένα απεσιόδοξο, ένα αισιόδοξο και ένα μετριοπαθές σενάριο. Για να σας δώσω μερικά μόνο στοιχεία, θα ήθελα να πω ότι αναμένουν ότι αν υπάρξει μια επιτάχυση της ανάπτυξης πολιτικών που θα εξασφαλίσουν την επίτευξη του στόχου του 20% των ανάσχημων πηγών ενέργειας ε, στην Ευρώπη 2020 το 2020 η ανάπτυξη της απασχόλησης θα είναι 2,76 εκατομμύρια θέσεις και οι εξαγωγές θα είναι 2,80 εκατομμύρια. Um, thank Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και αυτή την επικοδομητική συζήτηση και περιμένω με ανεπιμονησία την συνέχιση αυτής της συζήτησης. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Σλέμιγκερ. Äh, Θα σας απαντήσω σύντομα. Πολλά από όσα ανέφεραν εδώ οι σκιώδεις συζητητές με βρίσκουν σύμφωνοι. όσα είπε ο κύριος Λούντβινσον, ε, πραγματικά πηχούν τη δική μου σκέψη, δηλαδή θα πρέπει να υπάρξουν σταθερές ε, ε, συνθήκες επένδυσης των επιχειρήσεων. Αυτό θα είναι όφελος των εργαζομένων και της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης. Στη Γερμανία ε, γίνεται μια προσπάθεια αξιοποίηση των ανώσιμων πηγών ενέργειας. Και με αυτό συνδέω μετά όσα είπε η Κομισιόν. Θέλουμε να έχουμε μια πιο ανταγωνιστική Ευρώπη. Ναι, ακριβώ. Γι' αυτό θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τι εξαγωγέ. Και όσον αφορά του αριθμού που αναφέρεται στο τέλο, ε, μου προκαλούν κάποια θυμηδία. Αυτό δεν ισχύει μόνο στη Γερμανία. Ε, είμαι πεπισμένη ότι οι εξαγωγικές θέσεις εργασίας μπορούν να δημιουργηθούν όχι μόνο στην Γερμανία αλλά και σε άλλε χώρε, στην Ισπανία κλπ. Ότι οι εξαγωγέ δηλαδή δημιουργούν νέε θέσει απασχόληση. Δεν ισχύει μόνο για τη Γερμανία αλλά και για άλλε χώρε. Ε, κύριε Λούτφινσεν, έχετε δίκιο. Ε, δεν ε, θέλουμε μόνο θέσει απασχόληση υψηλών αποδοχών αλλά και στα χαμηλότερα και μεσαία επίπεδα και πραγματικά θεωρώ ότι είναι κυρίως ο τομέας ε, των χαμηλών αποδοχών όπου θα υπάρξουν οι μεταβολές και όπου θα πρέπει να αναπτυχθούν οι νέες δεξιότητες γιατί εδώ βρίσκεται το μέγιστο δυναμικό, το μεγαλύτερο δυναμικό. Στο μοντέλο Ευρώπη 2020 θεωρώ ότι αυτό δεν λαμβάνεται παρκώς ε, υπόψη. Το ξαναλέω, δεν πρόκειται για το τομέα των πανεπιστημίων, αλλά της ε, επαγγελματική κατάρτισης. Ε, εκεί θα πρέπει να δώσουμε την έμφαση. Και λέω προς την Επιτροπή ότι θα πρέπει να κοιτάξετε πιο προσεκτικά τις μελέτες που έχουν γίνει, τις διαβάσετε πιο προσεκτικά, να δείτε πού ακριβώς ε, εντοπίζετε το δυναμικό και να προσανατολίσετε εκεί τη μελλοντική σας στρατηγική, διότι νομίζω ότι αυτή την προοπτική έχουν υιοθετήσει και οι περισσότεροι συνάδελφοι εδώ στο σώμα. Τώρα, το ερώτημα το οποίο θέσατε εσείς, Ε, θα ήθελα να σε πιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι μια γρήγορη εξέλιξη διαφόρων ε, κλάδων εγκυμονεί επίσης κάποιους κινδύνους. Και όταν λέμε ότι θέλουμε να αξιοποιήσουμε το δυναμικό των θέσεων απασχόλησης για να μπορέσουμε να ξαναδώσουμε τους ανθρώπους στην επιστήμη ότι μπορούν να ζήσουν από αυτές τις ε, θέσεις απασχόλησης ε, νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει για παράδειγμα στον τομέα της ηλιακής ε, ενέργειας. Έχω διαβάσει τις σχετικές έρευνες. Πώς μπορούμε να συνδυάσουμε καλή εργασία και υψηλή ευελιξία. Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο θα πρέπει να θέσουμε στους κοινωνικούς εταίρους. Όχι μόνο στα συνδικάτα, αλλά και στα συνδικάτα. Δηλαδή, πώς μπορούν να συνεργαστούν. Αυτό ναι μεν πετυχαίνει στη Φιλανδία, σας πιστεύω απολύτως, 100% αλλά σε άλλε χώρε αυτό είναι δύσκολο. Και αυτό το λέω γιατί δεν θέλω ε, να παρουσιάσω τα πράγματα ρόδινα, αλλά θα ήθελα να εντοπίσω τα προβλήματα εκεί όπου ε, χρειαζόμαστε κατεπηγόντως την ανάληψη πολιτικής δράσης. Κατά τα άλλα θα ήθελα να σας ε, ευχαριστήσω Ε, έχετε κι εσείς μία έρευνα για αυτό το θέμα, μία μικρή σύνοψη, εάν θέλετε να εμβαθύνετε σε αυτή την προβληματική. Είναι αλήθεια, όπως είπε η Κομωσιόν, ότι σε αυτή την έκθεση απασχόληση 2009, στο παράρτημα αναφέρονται πάρα πολλές έρευνες που πραγματικά είναι αξιόλογες. Εγώ ίδια τις κοίταξα όλες και τις αξιολόγησα. Θεωρώ ότι επικύλουν ως προς την ποιότητά τους και τα συμπεράσματά τους, αλλά αν κάποιος θέλει να εμβαθύνει στο θέμα αυτό, ε, πραγματικά υπάρχει μια πληθώρα ε, προσεγγίσεων και στοιχείων και όλη η βιβλιογραφία που έχει συνοψίσει η Κομισιόν. Τώρα, το χρονοδιάγραμμά μας προβλέπει τα εξής. Ε, η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι στις 18 Μαΐου. Ε, δεν είναι τόσο πολύ καιρό ως τότε. Εγώ παρακαλώ τους σκιώδες συζητητές να έρθουν σε επαφή μαζί μου, για παράδειγμα Σύνοδο της Ολομέλειας, ε, να με ρωτήσουν που βασίστηκα, σε ποιες έρευνες στηρίζομαι κλπ. Ανά βάση στιγμή, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί μου. Η εισήτηση για τις τροπολογίες είναι στις 22 και 23 Ιουνίου στη συνεδρίασή μας. Η ψηφοφορία θα γίνει στις 13 και 14 Ιουλίου και μετά τη θερινή πάυση, μάλλον στην πρώτη Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου, αλλά ενδεχομένως και στη δεύτερη Σύνοδο ολομελία. Είναι σημαντικό ότι το αργότερο στη δεύτερη Σύνοδο του Ολομελίου ε, της Ολομελίας, συγγνώμη, η Βελγική Προεδρία ε, δίνει μια προτεραιότητα σε ζητήματα της αγοράς εργασίας. Και στη συνέχεια θα διοργανωθεί μια συνδιάσκεψη γι αυτό, για, τα, για εργασιακά ζητήματα. Ε, γι' αυτό θέλουμε προηγουμένως να έχουμε καταλήξει σε μια θέση ως προς την έκθεσή μας. και φανταζόμαστε ότι συνέχεια θα πάει στο Συμβούλιο και το Δεκέμβριο θα υπάρξει σχετική απόφαση από το Συμβούλιο. Και έτσι εμείς ως Κοινοβούλιο, οι συντονιστές που συμπεριλάβαμε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη, δίνουμε το έναυσμα για μια ανάληψη πρωτοβουλίας εκ μέρους της Επιτροπής. Τώρα, πότε θα συναντηθούμε, τη Δευτέρα 17 Μαΐου στο Στρασβούργο σε μια έκτακτη συνεδρίαση ε, στις 7 το βράδυ. Και η επόμενη συνεδρίαση είναι την 1η Ιουνίου, την 5η, στις Βρυξέλλες. Ε, στις 9 το πρωί έχουμε όλη τη μέρα μπροστά μας και το ίδιο ισχύει και για την Παρασκευή 2 Ιουνίου. Ε, με αυτές τις πληροφορίες θα ήθελα να κλείσω τη συνεδρίαση και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους παρέμειναν μέχρι το πέρας αυτής της συνεδρίασης για την υπομονή τους. Ευχαριστώ πολύ.